Good afternoon, colleagues. Um, welcome back and Χαίρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε και καλή χρονιά σε όλου. Ξεκινώ τη συνεδρίαση με την έγκριση τη ημερησία διάταξη. Σημεία 4 έω 14. Εξέταση γνωμοδοτήσεων για την απαλλαγή 2016 που αναβάλλονται για τη συνεδρίαση Σιλίμπε τη 14 η Ιανουαρίου. Και αυτή είναι η μόνη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη όπω τροποποιήθηκε. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχουμε μόνο ένα θέμα στην ημερήσια μα διάταξη. Θα επικεντρωθούμε στι προτεραιότητες τη Ολλανδική Προεδρία. Πρέπει να σας αναφέρω και τις γλώσσες. Δεν έχουμε κροατικά, λετονικά και ε, κελτικά στη διερμηνία μας και ζητώ συγγνώμη επίσης πρέπει να αναφέρω και την έγκριση των ε, αποφάσεων των συντονιστών πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση με την ε, Προεδρία. Έχουμε τους, τους συντονιστές και τις αποφάσεις με βάση το άρθρο 205 του κανονισμού. Η κυρία Χολμάιερ ονομάζεται, ορίζεται ως εισηγήτρια για την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και την αντικατάσταση τη ε, ε, οδηγία πλαισίου του Συμβουλίου 2002-475 για την καταπολέμηση τρομοκρατία. Ε, οι συστάσει των συντονιστών είναι στη διάθεσή σα. Εγκρίνονται, ελπίζω. Ναι, και άρα περνάμε στο μοναδικό θέμα τη ημερησία μα διάταξης για σήμερα και προτείνω αγαπητοί συνάδελφοι να σταματήσουμε στις 5 το απόγευμα. Σήμερα προβλέπεται η συνεδρία των συντονιστών στις 5.30. Δεν τους βλέπω όλους τους συντονιστές μας σήμερα εδώ βέβαια. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εάν μπορούμε να φέρουμε πιο μπροστά τη συνεδρίες και των συντονιστών, για τις 5 δηλαδή. Εκτός βέβαια και αν ξεπεράσουμε το χρόνο μας. Αλλά ο, ο κύριος πρέπει να, πάει στις 5, να φύγει στις 5 παρατάτω για να πάει στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Άρα θα κοιτάξουμε να οργανώσουμε το χρόνο μας κατά αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Φανταστέρ, λοιπόν, Υπουργός ε, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και ο κύριος Κλάς Ντάικχοφ, Υφυπουργό για την Ασφάλεια και τη Δικαιοσύνη και Υπουργό Μετανάστευσης είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Τους καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά. Χαίρομαι που είστε εδώ στις Βρυξέλλες για να μα παρουσιάσετε τι προτεραιότητε τη Ολλανδική Προεδρία στα θέματα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών και θα πρέπει να καλωσορίσω βέβαια όλη την ομάδα της ε, Ολλανδική Προεδρία εκ μέρου των συναδέλφων και να πω ότι ε, προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή συνεργασία και παραγωγική συνεργασία στο επόμενο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι. Και προτείνω προς τους υπουργούς μας να μας κάνουν ε, ο καθένας την παρουσίασή του επί 10 λεπτά περίπου και να ακούσουμε στη συνέχεια τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις συντονιστών και βουλευτών. Θα έχουμε όμως αρκετό χρόνο, όπως είπα, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ξεκινώ με την παρουσίαση του κύριου Άρτη Φαντεστόρη, Υπουργού ε, θεμάτων, για θέματα ασφαλείας και δικαιοσύνης. Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη στηρίζεται στην παράδοση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και, της... και των δικαιωμάτων. Πρόκειται για τις αρχές του κράτους δικαίου και δεν αφορούν μόνο Γάλλους, Γερμανούς, Έλληνες, αλλά όλους τους Ευρωπαίους και αν υπάρχει ένας υπουργός που να αντιλαμβάνεται τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ο υπουργός ή υπουργή των, για θέματα δικαιοσύνης και ασφάλειας στις τωρινές μας εποχές, τα θέματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ο Σάλφος Ντέικχοφ ε, θα σας απαντήσει στις ερωτήσεις σας τις σχετικές με τη μετανάστευση. Εγώ θα επικεντρωθώ στα θέματα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών. Αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι είναι ζωτική σημασία να συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω ήδη ε, τη χαρά να συναντήσω μέλη του Κοινοβουλίου σας ε, από τις επαφές μου στις Βρυξέλλες του Στρασβούργο τον προηγούμενο χρόνο. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ακρογωνιαία ηλίθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί το ένα όργανο να λειτουργήσει χωρίς το άλλο και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας εκθέσω τις προτεραιότητες του Συμβουλίου για την Ολλανδική Προεδρία. Ξεκινώ με τις εκκρεμότητες που θεωρεί σημαντικές το Συμβούλιο και θα ολοκληρώσω με θέματα ιστορικών, ε, ελευθεριών και δικαιοσύνης που θα δώσουμε εμείς έμφαση κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Θα αναμένεται ασφαλώς ε, αυτό που θα πω, ότι δηλαδή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ρουσπαστικοποίησης είναι στο επίκεντρο των ε, προσπαθειών μας και πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που κόστησαν τόσες ζωές στα κράτη-μέλη μας και θα ήθελα να απευθύνω θερμά συλληπιτήρια προς όλα τα κράτη αυτά και ιδιαίτερα στη Γαλλία η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να δώσει τις απαντήσεις, πρέπει πάντοτε να προσχωρούμε με τρόπο ισορροπημένο την προστασία δηλαδή του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως την προστασία του ιδιωτικού βίου, αλλά και ταυτόχρονα την ε, δίωξη, πάταξη και τιμώρηση των τρομοκρατών. Πρόκειται για μια ισορροπία λοιπόν και τα δύο στοιχεία πρέπει να προχωρούν ταυτόχρονα. Με τις πρόσφατες ε, επιθέσεις στο Παρίσι επιταχύνεται η επεξεργασία διαφόρων προτάσεων για την ε, καταπολέμηση δημοκρατία ή παραδείγματι και των πυροβόλων όπλων όπου θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις και ταυτόχρονα προτάσεις για το ποινικά μητρό. Είναι πολύ σημαντικά τα βήματα αυτά. Η οδηγία για την τρομοκρατία θα ενισχύσει τη δυνατότητά μα να καταπολεμούμε την τρομοκρατία. Θα καθιστά ποινικό αδίκημα τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, την ε, ε, εκπαίδευση σε τρομοκρατικέ δραστηριότητε ή την μετάβαση σε άλλο κράτο για την εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Και αυτά θα είναι βέβαια κύριε προτεραιότητε τη Προεδρία μα. Χαίρομαι που έχει εξασφαλιστεί συμβαστική λύση για την ε, καταγραφή των μητρών. Ευχαριστώ τον κύριο Κίρκοπ και όλους τους ε, συνεισηγητές για την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα στην ε, επεξεργασία των θεμάτων αυτών. Η οδηγία PNR λοιπόν για τα ονόματα επιβατών πτήσεων ε, θα προχωρήσει το χειρότερο δυνατό. Ιδιαίτερα δεν θέλω να αναφερθώ στους κύριους Άλμπρεχτ και Ορίστιμ για την, για την προσπάθειά τους στην οδηγία τη σχετική με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής αλλά ε, και νωρίτερα της Λουξεμβουριανής Προεδρίας είχαμε πολύ καλή συνεργασία και θα έχουμε πολύ καλύτερη προστασία στην ψηφιακή αγορά των προσωπικών δεδομένων. Σε συνεργασία μας θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το νομοθετικό πακέτο και μετά έχουμε την ε, εσωτερική στρατηγική για την ασφάλεια 2015-2020, ανανεωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική που θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά στις ε, απειλές θα, ε, και την άμυνα. Θα επικεντρωθεί σε αυτά λοιπόν η Ολλανδική Προεδρία με κοινέ δράσεις κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δουλειά της, Ολλανδικής, της Προεδρίας θα βρει συνέχιση και από την Ολλανδική αλλά στη συνέχεια και τη Σλοβενία και την Κυπριακή και την Μαλτέζικη Προεδρία. Με την 3 ε, 3 λοιπόν αυτή, η οποία βεβαίως θα συνεργάζεται πάντα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι μας θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στις δικές σας θέσεις. Θα συνεχίσουμε ταυτόχρονα και το τρέχον νομοθετικό μας πρόγραμμα και το σχετικό ιδιαίτερο με τις προτάσεις για, το για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και αξιόλογη δουλειά η Λουξεμβουριανή Προεδρία εν προκειμένου και θα συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή ως Ολλανδική Προεδρία. Η Λουξεμβουριανή Προεδρία έχει καταφέρει να κλείσει σχεδόν όλα τα άρθρα στα πρώτα πέντε κεφάλαια με τις κύριες διατάξεις για την οργάνωση της εισαγγελία, αλλά και τους κανόνες για, τις, για τη διερεύνηση της ανακρίσης και τις δημοσιονομικές ε, δικλίδες ασφαλείας. Πάνω στα επιτεύγματα αυτά θα στηριχθεί και η Ολλανδική Προεδρία, κλείνοντας προσωρινά τα ε, υφιστάμενα, τα εκκρεμή ακόμη κεφάλαια και προχωρώντας σε συνεργασία με τους εταίρους σημειώσω επίσης ότι λαμβάνουμε υπόψη όλες τις προτάσεις για το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την κυρία Ματέρα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, την συγκεκριά σας. Η πρώτη ομάδα εργασίας σήμερα ξεκινάει την επεξεργασία των άρθρων 56 έως 61. Η Προεδρία λοιπόν δείχνει ότι μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα και όλα στη δουλειά. Και έχουμε την οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με τα οικονομικά συμφερόντα της Ευρωπαϊκής ε, ε, των ευρωπαϊκών συμφερόντων, λεγόμενη οδηγία PAF. Είναι πολλά ζητήματα ακόμη αμφιλεγόμενα. Η Ολλανδική Προεδρία προσπαθεί να συνεχίσει, σκοπεύει να συνεχίσει τι συζητήσει ε, στο Συμβούλιο που είχε ξεκινήσει η Λουξεμβουργιανή Προεδρία με την ανάλυση όλων των σχετικών πτυχών και τη αρμοδιότητα ιδιαίτερα για τη δίωξη των ποινικών αυτών αδικημάτων με, στόχο να εξασφαλίσουμε αποδεκτές συμβαστικέ λύσει για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο υπό τη Λουξεμβουριανή Προεδρία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξασφαλίστηκε συμφωνία ως προς την οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας. Η κυρία Γκίσπερ και συγγήτρια και η κυρία Κινίτσι επίσης ε, αξίζουν συγχαρητηρίων για τις προσπάθειές τους για την ε, δικαστική αρρωγή, μάλλον για την ε, για το δικαίωμα της ε, νομικής αρρωγής ε, θα γίνει ακόμη προσπάθεια. Θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας ε, προτάσεις για την δικαιοδοσία ως προς τον κυβερνοχώρο, ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί διεξοδικά και θέλουμε να ενθαρρύνουμε την περαιτέρω συζήτηση του θέματος αυτού. Θα καταγράψουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το μέγιστο δυνατό φάσμα αρμοδιοτήτων και θεμάτων μπορεί να καλύψει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενδεχομένως προτείνοντας και νέα νομοθετήματα και λύσεις και σε σχέση με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Έχουμε αρκετά καλή βάση από τη Λουξεμβουριανή Προεδρία πάνω στην οποία θα στηριχθούμε. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα ζητήματα, κυρίε και κύριοι, που θέλει να υπογραμμίσει ιδιαίτερα η Ολλανδική Προεδρία. Μέσα σε μια διευρυνόμενη διαρκώ ψηφιακή αγορά έχουμε τεράστια δυνατότητα να αναπτύξουμε οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Άρα θέλουμε να ενισχύσουμε και την πρόληψη και την συνεργασία και την ασφάλεια και βέβαια τις, να προαγάγουμε τις, ιδιωτικές, τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα όπου ε, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη δύναμη σε σχέση με την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος μέσα από το κυβερνοχώρο. Η πολυτομιακή λοιπόν συνεργασία και η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών θα έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα για μας. Έχουμε προβλέψει τη διοργάνωση διασκέψεων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, ιδιαίτερα σε σχέση με το λαθρεμπόριο βάρος ανθρώπων, την ε, λαθροδιακίνηση μεταναστών και γενικότερα την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα να πω για ένα ζήτημα το οποίο ιδιαίτερα ενδιαφέρει τη δική σας Επιτροπή τα εξή. Ε, το κράτος δικαίου δεν είναι μόνο μία ε, αξία ε, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ένα εργαλείο για την προεγωγή της συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και έτσι έχουμε θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό ετήσιο διάλογο μεταξύ κρατών μελών για το κράτος δικαίου. 17 Νοεμβρίου του 2015 έγινε η πρώτη συνεδρίαση υπό τη Λουξεμβουριανή Προεδρία, η δεύτερη συζήτηση ε, υπό την Ολλανδική με τον Υπουργό Κούνερ των Εξωτερικών προβλέπεται για το Μάιο του 2016. Εν προκειμένου λοιπόν θα προσπαθήσουμε να στηριχθούμε πάλι στις επιτυχίες Λουξεμβουριανής Προεδρίας για να προχωρήσουμε και στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό προβλέπεται από τις συνθήκες. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνασα υπογραμμίζοντας την σημασία της ευρωπαϊκής ε, συνεργασίας. Και εδώ θέλω να συνεχίσω και τον διάλογο για το επόμενο εξάμεινο. Προσβλέπω λοιπόν σε πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Είμαι στον Υπουργό Ντάικοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ε, χαίρομαι και εγώ που σήμερα με προσκαλέσατε στη σημερινή συνεδρίαση για μια ανταλλαγή απόψεων, κυρίως σε σχέση με τη μετανάστευση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για τα κράτη-μέλη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό τη και τα αποτελέσματα που μπορούν να έχουν τα σημερινά φαινόμενα αν δεν καταλήξουμε σε ικανοποιητικέ λύσει. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που ε, έρχομαι σήμερα διότι σε αυτό το τομέα όλος ιδιαιτέρως ε, κρίνω ότι είναι μονόδρομος η συνεργασία. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα κράτος μέλος μόνο του ή ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει τη λύση. Ε, είναι κεντρική σημασία λοιπόν η συνεργασία ε, και δεν μιλώ για το Συμβούλιο, θα πρέπει να είμαστε και λίγο μετριοπαθείς. Ε, φυσικά χρειάζεται συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά οπωσδήποτε ε, χρειάζεται συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε στα πλαίσια του επιμερισμού των καθηκόντων και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, βιώνουμε μία προσφυγική κρίση, μία βαθιά κρίση Βλέπουμε όλοι τις εικόνες, δεν χρειάζονται καν λέξεις. Μπορείτε να κλείσετε τις εφημερίδες, να κλείσετε τον υπολογιστή ή την τηλεόρασή σας. Ορισμένες φορές είναι μεγάλη, μεγάλος ο πειρασμός για να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία, γιατί είναι φρικτές οι εικόνες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ε, εκλείπουν τα φαινόμενα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ένα θεσμικό επίπεδο ή σε κοινωνικό επίπεδο αυτά είναι πραγματικά ζητήματα, υποφέρουν καθημερινά οι άνθρωποι στο μέτρο που εμεί δεν μπορούμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση και είναι αμφίδρομη διαδικασία. Θέλουν μια καλύτερη ζωή, αυτό είναι το κινητρό τους ε, και ε, πέφτουν στα χέρια, πέφτουν θύματα αμήλικτων ε, διακινητών και σε υπερφορτωμένα σκαφίδια προσπαθούν να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Ε, υπάρχουν αυτοί που δικαιούνται το καθεστώς ε, του πρόσφυγα και χρειάζονται τη βοήθειά μας, όμως ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε αυστηροί με όσους δεν το δικαιούνται και θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι είναι ανθρωπιστική σε φύση η συμπόνια μα, δηλαδή αυτοί που διώκονται και προσπαθούν να ξεφύγουν, να σώσουν τη ζωή τους και δικαιούνται το καθεστώ του πρόσφυγα, δεν μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία με αυτούς που δεν το δικαιούνται. Ουδέλω θα είχαμε υπερβολική πίεση στην κοινωνία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μια κρατέα συνεργασία, μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη στρατηγική ε, να αντιμετωπίσουμε τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης ε, και φυσικά θα πρέπει να έχουμε πιο σύγχρονα μοντέλα για την υποδοχή και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας νωρίτερα, ανάντι, δηλαδή στις χώρες από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες και από τις χώρες από τις οποίες προσπαθούν να ξεφύγουν. Επίσης, ε, θα πρέπει να ε, δείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου επί των προσφυγικών ροών, ότι κάνουμε αυτό που κρίνουμε εμείς ε, σωστό, ταυτόχρονα όμως να, δώσουμε, να υπάρξει και μια ανταπόκριση για τα θεμητά δικαιώματα και τις θεμητές προσδοκίες των πολιτών που καλούνται να υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους Ε, διότι ε, μην ξεχνάμε ότι ε, υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις κυβερνήσεις και αυτό ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να αναβάλουμε τη διαδικασία, μπορούμε να μετακυλήσουμε την ευθύνη, αλλά σε καμία περίπτωση μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δέχουμε την αισθανόμαστε αυτή την πίεση πολύ έντονα και γι' αυτό θέλουμε να εντείνουμε τη συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο το ταχύτερο δυνατό, το νωρίτερο δυνατό δυνατό στην όλη διαδικασία να δίνουμε απαντήσεις, απαντήσεις που χρειάζεται. Επίσης, πέρα από την τωρινή κρίση, πρέπει να προετοιμαστούμε και για το μέλλον. Δεν θα ε, διεκπαιρεωθεί το ζήτημα μέσα σε ένα χρόνο. Για να είμαστε ρεαλιστές ε, και να δώσουμε πιστικές λύσεις, ε, θα πρέπει να λειτουργήσουμε μακροπρόθεσμα. Δοκιμάζεται το σύστημα Σέγγεν με την προσφυγική κρίση. Το σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων δεν λειτουργεί όπως το θέλαμε, όπως το είχαμε φανταστεί, γιατί βασιζόμαστε πολύ στο κεκτημένο του, του κανονισμού του Δουβλίνου Δηλαδή διαχειριζόμαστε την εισρωή, όμως στη συνέχεια η μεταχείριση δεν δείχνει ότι ε, ελέγχουμε ε, την ροή και αυτό ε, πλήττει την αξιοπιστία, αν θέλετε, στα μάτια των πολιτών και σε πολλές περιπτώσεις, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά θέλω να μην πω ότι είναι ρεαλιστικέ αυτές οι εκτιμήσει ή ότι βασίζονται σε γεγονότα, αλλά τουλάχιστον εκείνοι βλέπουν τι συνέπειε. εκείνοι το νιώθουν καθημερινά, νιώθουν καθημερινά ποιες είναι οι επιπτώσει. Ε, αυτών των αποφάσεων, ε, διότι εμείς ε, οι θύνοντες θα πρέπει να αποδείξουμε στους ανθρώπους ότι έχουμε τον έλεγχο, να αποδείξουμε στους συμπολίτες μας ότι μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Είναι θεμητές αυτές οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα κυρίως μακροπρόθεσμα του συστήματος. Δεν υπάρχει τώρα η δανεική λύση, δεν υπάρχει ένας κατάλογος μέτρος που θα λύσουν όλα τα προβλήματα, ούτε νυχθημερών μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, ε, ούτε και βραχυπρόθεσμα. Όμως αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε παράλυση ε, ούτε πρέπει να χανόμαστε σε βαθιστόχαστες ε, αναλύσεις θα πρέπει για τα συμπεφωνημένα ήδη να δράσουμε, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μήνυμα της Προεδρίας μας. Θέλουμε να φέρουμε αποτελέσματα και σταδιακά να δείξουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Ε, τους περασμένους μήνες ε, ασχοληθήκαμε επιχαρτούμε αυτή την άσκηση και σίγουρα όλοι ξέρουμε πως η εφαρμογή ε, χρειάζεται περισσότερη προσοχή και είναι πιο απαιτητική. Ε, για το μηχανισμό κατάσταση, Βερυπίν, έχουμε προς το παρόν αυτή την περιορισμένη ε, ομολογουμένως λύση. Χρειάστηκε λοιπόν χρόνος και θα ήθελα να παρεμπιπτόντως να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι Εσεί δεν χρειαστήκατε τόσο χρόνο όσο χρειάστηκαν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και είμαι και ποιητή όταν το λέω αυτό. Στο μέλλον λοιπόν, με τα νέα μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας, πιστεύω, ελπίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε και στην ίδια επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο, το ώστε αμελητή επιτόπου και όχι πλέον επιχάρτου να καταλήξουμε σε λύσεις για την εφαρμογή. Ποια είναι τα βασικά σημεία, τα hot spots, τα κέντρα υποδοχής ε, που θα ε, ε, συσταθούν, που θα δημιουργηθούν και το θέμα της μετεγκατάστασης. Πρέπει να αποφύγουμε τις συζητήσεις περί προτεραιοτήτων, ε, τι είναι πιο σημαντικό, τα hot spots ή κατάσταση ε, Βλέποντας και κάνοντας, ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τι θα γίνει με την καταγραφή στην πρώτη χώρα υποδοχής. Αυτό είναι ένα σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την κατάσταση και έλεγχος της ροής. Τι σημαίνει αυτό. Αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις υποδοχής, ούτως ώστε να επιστρέφονται άμεσα αυτοί που δεν δικαιούνται προστασία ή το καθεστώς του πρόσφυγα, ώστε να καταπολεμήσουμε τη λαθρεμπορία και τη διακίνηση. Ε, φυσικά υπάρχει το θέμα της του Σέγγεν, η συμφωνία του Δουβλίνου που έχουμε και επί της οποίας θα γίνει ε, διεξοδική συζήτηση, διότι δοκιμάζεται το σύστημα από ε, τους ψηλούς αριθμούς προσφύγων. Δεν είναι ρεαλιστικές συμφωνίες που έχουμε, δεν ε, λειτουργούν εύρυθμα και σε κάθε περίπτωση ε, ε, ήταν καταδικασμένες η αποτυχία αυτές οι αποφάσεις. αν λέμε ότι μόνο η πρώτη χώρα υποδοχής πρέπει να, να αναλαμβάνει αυτούς τους ανθρώπους και οι υπόλοιπε δεν φέρνουν καμία ευθύνη, δηλαδή μια πολύ περιοριστική ερμηνεία του Δουβλίνου, καταλαβαίνουμε μια τέτοια ερμηνεία ερμηνεία είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. Βεβαίω, τα περισμένα χρόνια στην πράξη γινόντουσαν πολύ διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που είχαμε συμφωνήσει και τα δεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τόνισαν αυτό, διότι οι επιπτώσει. Ε, ε βιώνονται από τους ανθρώπους και βλέπουμε πόσο δοκιμάζεται το σύστημα. Δεν μπορούμε όμως να πετάξουμε στα σκουπίδια την, ε, τις συμφωνίες που έχουμε. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, θα πρέπει να υπάρξει σωστός επιμερισμός των ευθυνών και αλληλεγγύη ανάμεσα και στα θεσμικά όργανα αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη ώστε να δώσουμε ικανοποιητικότερες ερμηνείες των υφισταμένων συμφωνιών. Τώρα, ε, ανακοινώθηκε ότι έπεται ε, πρόταση τους επόμενους μήνες. Ε, φυσικά όταν μιλάμε για την ενίσχυση της, των λειτουργιών φύλαξης και διαχείριση των συνόρων, η Ολλανδική Προεδρία ανέλαβε τη δέσμευση να γίνει δήλωση περί αυτού του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Πρόεδρε, θα έρθουμε εγκαίρως ε, σε συνεννόηση για τους τριμερείς διαλόγους που θα χρειαστούν ε, επί τη βάση μιας ε, κοινή αντίληψης σε σχέση με τα επιδιωκόμενα. Λοιπόν, θα διακόψω τώρα γιατί υπερεύνει και το χρόνο μου από τον ενθουσιασμό μου. Θα δώσω το λόγο, υπερεύνει το χρόνο που μου αναλογούσε σε σχέση και με την παρουσίαση του συναδέλφου. Ήθελα μόνο να πω πως στα πλαίσια της συνήθους ε, νομοθετικής διαδικασίας ο στόχος είναι ε, ε, εγκαίρως να εντοπίσουμε τα δύσκολα σημεία, να ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ για να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και εμεί η πολιτική των κρατών μελών και εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσουμε πού θα επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε γέφυρες ούτως ώστε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικέ λύσεις που θα έχουν να καταληξουμε σε ικανοποιητικές λυσεις σημασία για το μέλλον των πολιτών αλλά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Τάικοφ. Σας ευχαριστούμε και τους δύο και γιατί τηρήσατε και το χρόνο σας. Και αυτό το λέω και για να σας προειδοποιήσω λίγο. Έχουμε ένα κατάλογο μιλωτών ε, σχεδόν όλων εκείνων που βρίσκονται στην αίθουσα. Διαπίστωσα ότι όχι, δεν σας έχει υπερφορτώσει το πρόγραμμα ήδη, είμαστε στην αρχή του εξαμήνου, αλλά έχετε κατανοήσει πόσο ε, μεγάλο είναι το θέμα της μετανάστασης και φυσικά σας ενδιαφέρει και το θέμα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας ε, όπως και εμάς, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν. Προτείνω λοιπόν, επειδή είναι εδώ και τα μέλη και ο Υπουργός Ντάικοφ αναφέρθηκε σε τριμερείς διαλόγους και στην προετοιμασία, Είδατε το τελευταίο εξάμεινο ε, τι κάνουν τα μέλη μας, ε, τι κάνει το προσωπικό μας ε, και τι κάναμε στους τρισμερίδες διαλόγους το τελευταίο εξάμεινο. Ε, είναι πολύ, ήταν πολύ καρποφόρο το προηγούμενο εξάμεινο, αλλά τώρα θα αρχίσει και η διαδικασία των ερωτήσεων για τα πάντα. Επομένως σας προειδοποιώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να τα ξαντλήσετε όλα. Μπορείτε να απαντήσετε και αργότερα. Να απαντήσετε ό,τι μπορείτε να απαντήσετε. Και ο έλεγχος για την ε, Προεδρία είναι να κάνετε ό,τι μπορείτε για την νομοθετική σκοπιά και από εκεί και πέρα να τα δούμε όλα σταδιακά. Ε, υπήρχε πρόοδος και με τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία και ελπίζω ε, να υπάρχει αντίστοιχη με την Ολλανδική Προεδρία. Ε, Νομίζω ότι σας προειδοποιώ επιματέω, αλλά θα δείτε τι θα γίνει και ακόμα ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους συντονιστές. Θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές, θα απαντήσουν. Είναι η Ολλανδική Προεδρία, θα είναι σύντομη ούτως ή άλλως, λακωνική. Ε, και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε όλα τα υπόλοιπα μέλη. Έχουμε άφθονο χρόνο στη διάθεσή μας. Στράβωσαν ήδη τα πράγματα γιατί δεν έχουμε συντονιστεί από το ΕΛΚ. Είναι κάποιο εδώ που να αντικαθιστά το συντονιστή. Αν έρθει κάποιο θα του δώσουμε το λόγο, αλλά θα ξεκινήσουμε με την Πυργιού Τσίπελ. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω την Προεδρία των Κάτω Χωρών. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη με τις ερωτήσεις μου. Η πρώτη με ερώτηση είναι αν υπάρχει κοινό ορισμός για το κυβερνοέγκλημα. Αν κάποιος ε, παίρνει όπλα ε, και κλέβει μια τράπεζα, τότε είναι η ληστεία τράπεζας. Αν κάποιος ε, κλέβει χρήματα από του λογαριασμού πέντε διαφορετικών ε, τραπεζών με ψηφιακά μέσα, τότε δεν είναι ληστεία τράπεζα, είναι κυβερνοέγκλημα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν είναι πάλι αυτό ληστεία τράπεζα, αλλά με διαφορετικά μέσα. Ε, έχουμε ορισμό του κυβερνοεγκλήματος, λοιπόν. και καταλαβαίνω γιατί μπορεί να χρειάζονται διαφορετικά μέτρα για να ε, ε, διαπιστώσουμε και να συλλάβουμε εγκληματίες αυτής της μορφής, αλλά ε, το θέμα είναι τι γίνεται με τη δίωξή τους από εκεί και πέρα. Τώρα, για την τρομοκρατία. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς Ευρώπης για να δούμε πώς κινούνται οι ροές χρημάτων, αλλά τι κάνετε εσείς, είστε σε επαφή με άλλους για να προσπαθήσετε να σταματήσετε ίσως την πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη στην τρομοκρατία ε, από χώρες ε, όπως η Τουρκία ή η Σαουδική Αραβία. Διότι αν δεν μπορέσουμε να τα σταματήσουμε εκεί, ίσως δεν αρκεί να σταματήσει η χρηματοοικονομική στήριξη από πλευράς Ευρώπης. Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, όπως διαπιστώνουμε την κατάσταση τώρα εδώ στην Ευρώπη, θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθούμε πολύ περισσότερο στη χρήση των μέσων που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο διάβασα στι εφημερίδε ότι ένας από τους δράστες ε, στο Παρίσι ε, ζούσε ε, παριστάνοντα τον πρόσφυγα σε διάφορες περιοχές Ευρώπης με διάφορα ονόματα. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς υπάρχει λοιπόν πρόβλημα στην καταγραφή και στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από όλου. διότι αν είχε γίνει αυτό θα είχαμε διαπιστώσει ότι το εν λόγω άτομο ήδη περιλαμβάνεται στο σύστημα με αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα αλλά με άλλο όνομα. Ε, ίσως λοιπόν υπάρχει πρόβλημα εκεί και ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε και σε αυτό και να μην αναφερόμαστε μόνο στο κλείσιμο των συνόρων μας ε, και στην απαγόρευση εισόδου για όλους όσον αφορά τη μετανάστευση. Ένα εξυγχρονισμένο μοντέλο ε, παροχής ασύλου. Συμφωνώ ότι και οι πρόσφυγες ε, χρειάζονται και αυτοί έναν ασφαλή χώρο στις χώρες καταγωγής τους και στις χώρες διέλευσης. Αλλά ε, ορισμένες φορές έχω την εντύπωση όταν παρακολουθώ τις συζητήσεις και δημοσίως αλλά και από πλευράς κυβερνήσεων προκύπτει ίσως ότι θα θέλαμε τους πρόσφυγες μόνο σε τρίτες χώρες. Ποιες είναι αυτές οι τρίτες χώρες, Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία, Πακιστά, αν αυτές είναι χώρες οι οποίες είναι πολύ φτωχότερες από πολλές από τις ευρωπαϊκές μας χώρες. Ε, πράγματι λοιπόν ο στόχος είναι να υπάρχουν πρόσφυγες μόνο εκεί. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό και δεν νομίζω ότι και εσείς θέλετε μια τέτοια απάντηση. Θεωρώ όμως ότι αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις τρίτες χώρες στον τομέα αυτό, θα πρέπει να αποτελέσουμε εμείς το καλό παράδειγμα για το πώς αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί, όχι μόνο όσον αφορά την υποδοχή και την καταγραφή τους, αλλά και όσον αφορά την ε, ε, μετεγκατάσταση, αλλά και την ένταξη των προσφύγων. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση τώρα Ε, στη ρίση που ακούμε συχνά ότι οι πολίτες μας δεν θέλουν πρόσφυγες. Βεβαίως και θα το πούν αυτό γιατί πολλοί πολιτικοί, πολλοί σημαντικοί παράγοντες αυτό δηλώνουν και ορισμένες φορές δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα ή κάποια κυβέρνηση η οποία να τους διαψεύδει. Ο κόσμο λοιπόν είναι απογοητευμένο, δεν βλέπει άλλη λύση και σαφώ ακολουθήσει αυτή την άγουσα. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη όμως πολιτική ηγεσία η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Και μια πάρα πολύ σύντομη παρατήρηση για τη Σέγγεν. Όσον αφορά τις ροές προσφύγων και την τρομοκρατία, πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τη Σέγγεν και να ξαναρχίσουμε ελέγχους σε όλα μας τα σύνορα. Καταρχάς, είμαι βέβαιη ότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθήσει ε, με το θέμα των προσφύγων και κατά δεύτερο, εάν κλείσουμε τα σύνορά μας ε, σε εθνικό επίπεδο, ε, σίγουρα αυτό δεν αποτελεί μόνο αρνητική λύση για τους πρόσφυγες, αλλά θα επηρεάσει αρνητικά και την οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη. Καλό θα ήταν λοιπόν να κάνουμε μια νέα αρχή και σας διαβεβαιώ ότι θα σας υποστηρίξουμε και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να εξεύρουμε μια λύση και να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό και εντό αλλά και εκτό Ευρώπη με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι είδαμε τον τελευταία χρονιά. Ευχαριστώ κύριο Κύρκοφ από πλευράς Ευρώπης Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Πρόκειται για μια χρονιά η οποία θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω την Ολλανδική Προεδρία και να καλωσορίσω και τους επικεφαλής ε, για τα θέματα τα οποία μας παρουσίασαν και θα ήθελα να σταθώ στα θέματα αυτά και μετά να σταθώ λίγο περισσότερο στη μετανάστευση και σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Καταρχά, το επιχείρημα το οποίο μα ανέφεραν ότι θέλουν να επικεντρωθούν στην ουσία και να υπάρξει μια προστιθέμενη αξία σε αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, φαίνεται μια πολύ λογική προσέγγιση και το γεγονό ότι επικεντρώνονται στη συνεργασία είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι απαραίτητο περισσότερο από ποτέ σήμερα λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ των κρατών μελών είναι ένας απαραίτητος ε, και επιθυμητός στόχος και φυσικά ευπρόσδεκτος και από εμάς. Χρειαζόμαστε τα μέτρα τα οποία θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, ικανούς ε, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις οικονομικές προκλήσεις αλλά και τις άλλες προκλήσεις που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά για θέματα ασφαλείας. Χαίρομαι λοιπόν για αυτά τη γενική θεματολογία που μας παρουσιάσατε και επίσης να σας πω εδώ ότι το γεγονός ότι η Ολλανδική Προεδρία θα συνεργαστεί και με τη Σλοβακία και με τη Μάλτα, τις δύο επόμενες προεδρίες δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας καθησυχάζει όλους και χαίρομαι που θα ε, συνδράμουν και αυτοί με τις ε, επόμενες προεδρίες και θα είναι πολύ καλό και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τις επόμενες προεδρίες. Να περάσω τώρα στο προκείμενο. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Δουβλίνο καταρχάς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Είμαστε στη διαδικασία εξέτασης της του Δουβλίνου πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός του διπλίνου που να το σέβονται όλα τα κρατημέλη. μελη Οτιδήποτε περιλαμβάνει ο κανονισμός θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Θα πρέπει ίσως να υπάρχει και μία σχέση μεταξύ της κατάστασης ε, συνόρων Σέγγεν ε, και των κρατών μελών και τη δυνατότητα ή την αδυναμία τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του. Δεν ξέρω αν η Προεδρία συμφωνεί ότι θα πρέπει να έχουμε σαφέστερου κανόνε ε, όσον αφορά ε, την προσπάθεια που επισημαίνει το Δουβλίνο. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω πιο συγκεκριμένα, ε, κύριε Πρόεδρε, είναι η ριζοσπαστικοποίηση. Νομίζω ότι πρόκειται για κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πολύ εμείς εδώ και στην Επιτροπή μας, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως και άλλοι έχουν πει, η ριζοσπαστικοποίηση είναι εσωτερικό ζήτημα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει κάτω από τα μάτια μας. Και εγώ πιστεύω ότι είμαι προσωπικά υπεύθυνο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι νομοθέτες θεωρούν ότι είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Ε, και φαντάζομαι ότι και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία. Το θέμα που με ενδιαφέρει πολύ, το γνωρίζετε, είναι να υπάρχουν νόμοι που να μας επιτρέπουν να συλλάβουμε τους δράστες ε, και να υπάρχουν κατάλληλες διώξεις. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση σε ολιστικό επίπεδο και να αντιμετωπίσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση στην πηγή της και όχι να κάνουμε όπως συνήθως τίνουμε να κάνουμε περισσότερα στο τέλος μιας διαδικασίας επειδή μας έχει δυσκολέψει. Ε, δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η Προεδρία προκειμένου να... Ε, αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τους. Αλλά ε, να πω ότι χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας συνδράβουμε και να συνεργαστούμε μαζί σας για το έργο σας. Η κυρία Βουίξτρομ από πλευράς Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ την Ολλανδική Προεδρία. Προσβλέπουμε στην συνεργασία μαζί σας και να τονίσω και εγώ αυτό το οποίο ακούστηκε, ότι αναλαμβάνεται τα ενία της Προεδρίας ε, σε μια στιγμή η οποία αποτελεί πρόκληση και είναι πολύ δύσκολη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε λοιπόν που, είμαστε, που είστε εδώ και προσβλέπουμε στη συνεργασία. Να σταθώ λοιπόν και σε κάποια θέματα στα οποία θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες κινήσει στη διάρκεια τη Προεδρίας σα. Στη διάρκεια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας ε, είδαμε ότι προσπάθησαν να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε μια ίση κατανομή για ένα δίκαιο σύστημα ε, επανεγκατάστασης. Μετεγκατάσταση, συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, τελευταία εβδομάδα αναφέρθηκε στο θέμα με την κατάσταση και πρέπει να πω ότι είναι απογοητευτικό και ε, αποτελεί κατάθλιψη να ακούμε τι δεσμεύσει αναλάβαμε. Και το αναφέρατε και εσεί, κύριε Υπουργέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδρασε πολύ γρήγορα. Ναι, εμεί ετοιμαστήκαμε σε τρει μέρε και το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Έχετε πολλή δουλειά λοιπόν να κάνετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε αυτή την πολύ καλή ομαδική εργασία την οποία μα επισημάνατε ω τόσο η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι θα κάνετε ώστε τα κράτη-μέλη να παραμείνουν σε μια διαδικασία όπου πραγματικά θα δεσμευθούν να συνεργαστούν και να συνεισφέρουν με δίκαιο τρόπο ώστε να υπάρξει πραγματική δράση στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης. Δεύτερον, για την ε, διαβόητη αυτή η νέα πρόταση για το Δουβλίνο. Λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε ανεπισήμως να ακολουθήσουμε μία ε, προσέγγιση ε, ελαχίστων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Δηλαδή να ακολουθούμε μόνο τις αποφάσεις του δικαστηρίου που σχετίζονται μόνο στους ε, ασυνόδευτους ανηλίκους. Δυστυχώ δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων και επομένω θα ήθελα να ξέρω εσεί τι σκοπεύετε να κάνετε ως Προεδρία για αυτό το ζήτημα το οποίο μπορεί να φαίνεται ίσονο σημασία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίση να πω ότι δεν θα μπορούσε να γίνεται ανταλλαγή απόψεων σήμερα αν δεν αναφέρω το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητούμε συνεχώς, αλλά γιατί αφορά τις βασικές αρχές επί των οποίων δράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι αξίες αυτή τη στιγμή ε, απειλούνται σε αρκετά κράτη-μέλη. Θα μπορούσα να αναφέρω και πάλι την Ουγγαρία και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφέρω και την Πολωνία. Αλλά υπάρχουν ανησυχητικές τάσεις και σε, άλλους, σε άλλα κράτη-μέλη. Η Ολλανδική Προεδρία σήμερα λοιπόν εξετάζει ίσως κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το θέμα αυτό, ώστε επιτέλους στην Ευρώπη το Συμβούλιο να απομακρυνθεί από αυτή την πολύ βολική πολιτική σιωπή ε, που, ε, στην οποία έχει παραμείνει ε, το τελευταίο διάστημα, ε, το οποίο δεν βοηθάει κανέναν, παρά μόνο αυτούς οι οποίοι υποσκάπτουν τις θεμελιώδεις αρχές ε, και το κράτος δικαίου. Θα ήθελα να δω αν επιτέλους θα υπάρξει κάποια προεδρία που θα είναι διατεθειμένη να κάνει κάποια κίνηση από αυτού, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Δίο από πλευράς ΚΟΕ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα αξιοποιήσω την ευκαιρία που έχω να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, το Ολλανδικά. Εύχομαι φυσικά καλώς ορίσατε στους Υπουργούς και κάθε επιτυχία στην Ολλανδική Προεδρία. Και ελπίζω ότι θα καταλήξουν σε καλά αποτελέσματα στους τομείς κρίσης που ανήκουν στις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής και βεβαίως το να εξευρεθεί λύση θα είναι προς το συμφέρον όλων μας. Είναι αυτονόητο αυτό. Θέλω όμως να προσθέσω το εξής. Η Προεδρία αυτή, και αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση, θέλει να δράσει με τρόπο ρεαλιστικό, πραγματιστικό όπως λέει. Με ένα όραμα που θέλει να υλοποιήσει. Όραμα που φαίνεται να λείπει σε ορισμένου τομεί. Και πρέπει να δείτε πώ θα βρείτε τι συμβαστικέ λύσει, αλλά ίσω δεν είναι αυτή το καλύτερο σημείο κίνηση. Οι κάτω χώρε ήταν ανέκαθεν η χώρα η οποία ε, προσυπέγραφε τις συμφωνίες σχετικές με τα προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν θα έπρεπε να είναι το έμβλημα της επόμενου, του επόμενου εξαμήνου σε πολλούς τομείς. Ο Υπουργό Φαντεστόρ επίση μα ανέφερε τη σημασία που αποδίδει στο κράτο δικαίου αλλά και οι διορισμοί δικαστών, επί παραδείγματι, έχουν μεγάλη σημασία σε αυτό, όταν λέγεται ότι πρέπει να υπάρχει διάλογο και με άλλους υπουργούς. Διερωτώ με. Διερωτώ με, τι θα πούμε στους Πολωνούς συναδέλφους και φίλους. Το κράτος δικαίου πρέπει να είναι μία από τις κυρίαρχες αρχές και πρέπει να είναι για το επόμενο εξάμεινο. Στους Πολωνούς λοιπόν συναδέλφους σας, τι θα λέγατε, γιατί και εγώ διερωτώ με αν ήμουν στην Προεδρία, τι θα έλεγα, ε, για την... Ε, δικαστική αρρωγή φαίνεται να αντιφέρεστε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση, μάλλον στην, ε, στο ευεργέτημα της παινίας φαίνεται να θέλετε να δώσετε έμφαση στη νομική δηλαδή αρρωγή στους ε, πιο αδύναμους, γιατί είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, αλλά θέλω να περάσω τώρα και στο θέμα των προσφύγων. γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο φαίνεται να μην μπορούμε να δώσουμε ε, εύκολα μακροπρόθεσμες λύσεις όπως ε, εκδηλώνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αλλά η κατάσταση είναι καταστροφική και αυτοί που υποφέρουν το περισσότερο είναι οι πρόσφυγες. Αυτοί υποφέρουν προς την τωρινή κατάσταση γιατί δεν βρίσκουν υποδοχή, δεν έχουν προοπτικές ε, για ταχεία διεκπαιρέωση της αίτησής τους σε οποιοδήποτε κράτος και να απευθύνονται στους πρόσφυγες και ακούω μάλιστα να αναφέρονται με κάποιες επιφυλάξεις τα θέματα των κέντρων υποδοχής, των hot spots. Εδώ δεν θέλω να πω ότι το ζήτημα της υποδοχής είναι ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί μακροπρόθεσμα. Εδώ πρέπει να γίνει σεβαστή η αξιοπρέπεια των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει αυτό να το επιδιώξουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα για την ανθρώπινο δικαίωμα. Και ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που θέλω να θέσω στον κύριο Ντέικοφ του Καλέ, αλλά και της Δουνκέρκης πλέον. Το Καλέ με 2.500 ανθρώπους που ζουν σε παραπήγματα, αλλά τώρα και στα περίχωρα της Δουνκέρκης, γιατί περιμένουν να βρουν ένα φορτηγό αυτοκίνητο στο οποίο θα επιβιβαστούν για να περάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα πρόβλημα το οποίο όμω βλέπουμε και στο Βέλγιο. Είναι γνωστό. Τι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε λοιπόν βράχει πρόθεσμα πρόκειται να αναλάβετε για να ε, υποχρεωθεί η Γαλλία να κάνει αυτό που οφείλει. Να τη πούμε δηλαδή ότι δεν μπορεί να αποστρέφει πλέον το βελέμα, πρέπει να χορηγηθεί το άσυλο και να χορηγηθούν, ε, να δοθούν οι λύσεις. Ιδάλλως πρέπει να ληφθούν μέτρα. Κυρία Σαρτζαντίνη, εκ μέρους των Πρασίνων. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους Υπουργούς. Κύριε Φαντεστόρ, κύριε Ντέικοφ, καλώς ήρθατε. Το Σταγματικό Δικαστήριο και η νομοθεσία στην Πολωνία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ο Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Ρούιτε ε, μίλησε με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα για το θέμα αυτό. Αλλά χρειάζεται και μια ηγετική ε, προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ντόναλτ Τούσκ, Πολωνός ο ίδιος, δεν είναι σε θέση να αναπτύξει αποτελεσματικά διάλογο με τον Πολωνό Πρωθυπουργό. Ελπίζω λοιπόν η Πολανδική Προεδρία να μπορέσουμε να ε, δούμε τα θέματα αυτά της Πολωνίας και του Σταγματικού Δικαστηρίου και να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις εγγύησεις που χρειάζονται για να καταπολεμηθούν ε, οι αντιδημοκρατικές αυτές τάσεις. Επίσης, σε σχέση με προτάσεις που τυπώσει η Ολλανδική κυβέρνηση πριν από την ανάληψη της Προεδρίας, τη δυνατότητα δηλαδή για περιορισμό των δυνατότητων μετακίνησης εκείνων οι οποίοι κηρύττουν το μίσος, περιορισμό της ελευθερίας διακίνησης εκείνων που υποστηρίζουν τη βία αυτό είναι μια πολύ σημαντική τοποθέτηση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι και στον Εμένο Βασίλειο που κάνουν τις δηλώσεις. Θεωρούνται και αυτοί ε, κήρυκες του μίσους. Θα ήθελα να μάθω ποιες θέσεις προβάλλει και υιοθετεί η Ολλανδική Προεδρία. Οι Γερμανοί δικαστές παλαιότερα, αλλά τώρα και οι Ολλανδοί δικαστές, λένε ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης πλέον δεν θα αποστέλουν κανέναν, ε, δεν θα εκδίδουν δηλαδή κανέναν κρατούμενο ή ύποπτο προς την Ουγγαρία. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με το άρθρο 3 της Συνθήκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ε, τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ε, γιατί υπάρχει κίνδυνος για απάνθρωπη αντιμετώπιση. Δεν θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να επανεξεταστεί ώστε με το ένταλμα ε, σύλληψης και την έκδοση να γίνονται σε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και κρατουμένων, η δυνατότητα πρόσβαση σε δικηγόρο και το καθεξής. Για δε την ασφάλεια και το έγκλημα. η Ολλανδική Προεδρία έχει προχωρήσει σε κάποια σκέψη σε σχέση με την περιγραφή της εσωτερικής κυβερνοασφάλειας. Γιατί έχετε κάνει πολλή δουλειά γενικά, αλλά για την εσωτερική κυβερνοασφάλεια δεν υπάρχει ορισμός ευρωπαϊκός ενιαίος. Αντιμετωπίζουμε διασυνοριακές απειλές και θα ήταν σκόπιμο να έχουμε ένα τέτοιο ορισμό και βέβαια θα ήθελα να ε, μάθω τις δικές σας θέσεις για τους πρόσφυγες τώρα και τη μετανάστευση. Χτες ακόμα στην Ολλανδική τηλεόραση, σε μια εκπομπή, ο Πρωθυπουργό των Κατοχωρών Χωρών, Ρούιτε, ε, επεσήμανε, σημείωσε ότι θα πρέπει οι κινήσεις της μετανάστευσης να φτάσουν σε μηδενικά επίπεδα και ότι για το στόχο αυτό είναι διότι βάλει σημαντικά ποσά στην Τουρκία. Αυτή είναι πράγματι η στόχευση της Ολλανδικής ε, κυβέρνησης και οι πληρωμέ αυτέ, τα ποσά που ακούγεται ότι θα είναι μέχρι και 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και τίποτα δεν έχει ακόμη καταβληθεί, πιστεύετε ότι θα αρκέσουν ώστε να συγκρατηθούν αυτέ οι μεταναστευτικέ ροέ. και ποιο θα πληρώσει τι, σε τι αναλογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση, στον, ε, στο θέμα της επανεγκατάστασης προσφύγων που βρίσκονται στην Ιταλία και την Ελλάδα. Εδώ και 1,5 μήνα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κάτω χώρες ότι οι 100 πρώτοι εκ των 1.500 υποψήφοι για μετεγκατάσταση θα πρέπει να φτάσουν 100 χώρες. Περισσότεροι από 1.500, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να είχαν ήδη επαναγκατασταθεί οι 100 πρώτοι. Τίποτα δεν έχει γίνει εδώ μεταξύ. Και βέβαια δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ιταλία και την Ελλάδα. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό ξέρουμε. Θα μας πείτε λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με τα hot spots και ποιοι είναι οι λόγοι που εξηγούν αυτά τα φαινόμενα. Δεν θα πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί όλοι πρέπει να δράσουμε από κοινού. Δεν αρκεί να μιλούμε μόνο, πρέπει να δράσουμε. Η Ολλανδική Προεδρία έχει συγκεκριμένες πρακτικές και πραγματιστικές, όπως λέτε, προτάσεις ε, για το θέμα αυτό. Κατά τη διάρκεια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, ε, κάποιες δεκάδες μόνο προσφύγων εγκαταστάθηκαν, ε, δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα και να γίνουν σεβαστές οι ποσοστώσεις όπως έχουν προβλεφθεί από τα κράτη-μέλη. Επίσης θέλω να ρωτήσω για έναν Ολλανδό Υπουργό, ο οποίος ακούστηκε να προτείνει σε μια πολιτική εκπομπή στην Ολλανδική τηλεόραση κάποιες ε, ε, ιδέες για ένα μίνι Σέγγεν και στην εκπομπή που ανέφερα νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Ρούτε και τελειώνω Πρόεδρε έλεγε ότι αν μέσα στους επόμενους μήνες δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των προσφύγων θα αναλάβουν μονομερή μέτρα οι κατοχώρες. Τι εννοείται ως μονομερή μέτρα. Αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας τους υπουργούς πέραν των συγκεκριμένων νομοθετικών προτάσεων, ε, τις οποίες σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε ε, εντατικά, θα πρέπει να εξετάσουμε ε, ιδιαίτερα τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, γιατί αυτό είναι ο σύνδεσμος για τα πάντα. Αυτό που λέω μπορεί να θεωρείται δεδομένο, αλλά είναι τόσο δεδομένο όσο και βασικό για να υπάρχει μία ε, συνεργασία μεταξύ ε, κρατών μελών, όταν δεν υπάρχει διάθεση για συνεργασία, δεν υπάρχει κάποιο μέσο που να μπορεί να ισχύει. Δεν υπάρχει κανονισμός ή οδηγία που να μπορεί να είναι χρήσιμο και να αποτελεί λύση για ένα πρόβλημα, όταν μετά δεν υπάρχει διάθεση για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και το διευκρινίζω αυτό με βάση και τα όσα διαπιστώσαμε να συμβαίνουν τελευταία. Ε, στη πλειοψηφία των περιπτώσεων κάθε πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομοθετική και η οποία είχε συζητηθεί με βάση κοινοτικού όρους έφτανε στο Συμβούλιο και εκεί ε, ε, την ε, κατακαιρματίζαμε και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση στο τέλος ε, έμενε κενή νοήματος. Το είδαμε και με τις πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι και την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπήρχε μια σαφής ε, δήλωση ότι υπήρχαν μεν πληροφορίε, αλλά δεν έγινε ανταλλαγή πληροφοριών. Και αυτό λόγω έλλειψη διάθεση συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είτε πρόκειται λοιπόν για τα πολέμηση τη τρομοκρατία, όπου πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να γίνουν πολλά, είτε πρόκειται για καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο, σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση, αλλά το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η διάθεση για συνεργασία. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε πόσο είμαστε διατεθειμένοι να συζητούμε σε κοινοτικού όρους και πόσο είμαστε διατεθειμένοι να συζητούμε σε διακυβερνητικούς όρους. Γιατί δάλλως, επαναλαμβάνω, θα μπορούσαμε να συζητάμε χιλιάδες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες θα είναι παντελώς άχρηστες αν δεν υπάρχει συνεργασία όσον αφορά τη μετανάστευση. Αναφερόμαστε σε σύστημα υποδοχή, αλλά πολύ συχνά δεν αξίζει να το αποκαλούμε σύστημα υποδοχή το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται. Πρόκειται για ένα αποτυχημένο σύστημα, το οποίο και πάλι ε, πλήττεται από έλλειψη συνεργασίας ε, και το σύστημα με την κατάσταση είναι αποτυχημένο. Τα ποσά, ε, οι αριθμοί που γνωρίζουμε μέχρι πρόσφατα ήταν 159 μόνοι μετανάστε οι οποίοι μετεγκαταστάθηκαν με, από του 160.000 ε, νομίζω ότι με αυτή τους ρυθμούς δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Είπατε κύριε Υπουργέ ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά τους ε, παράνομους μετανάστες και πρέπει να ενισχύσουμε τον επαναβατρισμό. Ωραία, αλλά πώς. Πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα που δυσκολεύεται να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναπατρισμού. Πώς μπορούμε να κάνουμε επαναπατρισμό με προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πώς μπορεί να γίνει επαναπατρισμό αν δεν υπάρχει διμερή συμφωνία. Ωραία, να τις βοηθήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες επαναπατρισμού, αλλά στην πράξη πώς θα την εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση. Και για τη Σέγγεν και πάλι. Πρέπει να την ξανασυζητήσουμε. Δεν λειτουργεί. Ε, τι σημαίνει να την ξανασυζητήσουμε τη Σέγγεν. Ή υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία ή δεν υπάρχει. Ε, η ενδιάμεση οδό θα μπορούσε να είναι μια μήνυ Σέγγεν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μα διευκρινίσετε. Αναφέρεστε πραγματικά σε μια μήνυ Σέγγεν. Τι σημαίνει αυτό, τι προποθέτει, ποιο θα την αποφασίσει και πώ θα εφαρμοστεί. Ιδάλω, επαναλαμβάνω, υπάρχει ή δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία. Εάν θα αποφασίσουμε να αμφισβητήσουμε τη Σέγγεν, σημαίνει ότι θα καταρρεύσει ένα από του πυλώνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε σκεφτεί τι συνέπειε θα μπορούσε να έχει αυτό για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Και τέλο, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου, συμφωνώ απολύτω. Ήμουν εισηγήτρια τη έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα για το 2013-2014 και διαπίστωσα πόσο μεγάλη δυσκολία υπήρχε στην εξέβρεση συνένεση, όσο το δυνατόν ε, με βάση την πλειοψηφία για την παρακολούθηση της κάθε χώρας. Σας ρωτώ λοιπόν τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να διασφαλίσουμε ότι θα γνωρίζουμε πραγματικά και θα λαμβάνουμε πληροφορίες για το κράτος δικαίου στην κάθε χώρα και αυτό με στόχο να κατανοήσουμε πραγματικά εάν και εφόσον πρέπει να παρέμβουμε και με ποιο τρόπο, ε, με προληπτικό τρόπο. Γιατί αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προλάβουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην δρούμε κατόπιν εορτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέτσολα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Κλοντ. Θα ήθελα κι εγώ, όπως και οι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ολλανδικής Προεδρίας για τις παρουσιάσεις που έκαναν. Είμαι από τη Μάλτα και Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, εν ώψη και της μελλοντική ε, προεδρίας, ε, να έχουμε μια ε, πολύ καλή συνεργασία με την Ολλανδική Προεδρία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με αυτό που ξεκίνησε πέρυσι αλλά και ευρύτερα από τις ε, τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές ε, και μετά. Συνεργάζομαι με την συνάδελφο Κάγκα και είμαι συγγήτρια για αυτό το ζήτημα. Τα θέματα θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, στο Στρασβούργο. Ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν πρόκειται να συζητήσουμε τον κανονισμό Δουβλίνου, αν πρόκειται να πραγματευτούμε όλα αυτά τα ζητήματα μετανάστευσης, θα πρέπει να αγγίξουμε και το θέμα της αλληλεγγύης, να συζητήσουμε διεξοδικότερα το θέμα της μετεκατάστασης. Τους τελευταίους έξι μήνες δεν έχουν γίνει πολλά στην πράξη. και καλώ την Ολλανδική Προεδρία να ασχοληθεί με ακριβώ αυτό το ζήτημα τη απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο του τελευταίου έξι μήνες. Το ΕΛΚΑ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θέλει να προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του δικαιώματος ασύλου, της εφαρμογής των κανονισμών, της ευθύνης των κρατών μελών ως προς την υλοποίηση των συμφωνιών που υπάρχουν. Θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στις χώρες για να εφαρμοστούν οι συμφωνίες, τα πρότυπα, η εφαρμοστή νομοθεσία γενικότερα που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Για τους συνοριοφύλακες Καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους επόμενους 6 μήνες φυσικά θα, θα αναδείξουμε σε προτεραιότητα αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος, θα ήθελα να ζητήσω από τους Υπουργούς ε, να σχολιάσουν ε, αυτές τις ε, παρεμβάσεις. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλους 13 συναδέλφους που θέλουν να παρεύουν, οπότε πρέπει να κρατήσουμε και λίγο χρόνο. Ε, όμως θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις διότι Σα απιθυνα συγκεκριμενε συγκεκριμένε ερωτήσεις. 5-6 λεπτά αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πω για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που σήμερα από πλευρά του Συμβουλίου μπορώ να συμμετάσχω στη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα τρομοκρατία. Θα είναι προτεραιότητα για μας η εφαρμογή των επιχειρησιακών μέτρων σε σχέση με την αναθεωρημένη ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια, κυρίως ως προς την ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως εξάλλου ανέφεραν και οι βουλευτές. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα για το επικείμενο άτυπο συμβούλιο και χαιρόμαστε φυσικά που θα εκπροσωπηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πώς να εξασφαλίσουμε την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών και δεύτερον η εφαρμογή ε, των συμφωνιών μας και κυρίως ε, του PNR για τα στοιχεία επιβατών. Πρέπει να προστατεύσουμε ε, το κοινό από τις επικείμενες απειλές, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τα βασικά δικαιώματα. Είναι λεπτή ισορροπία. Κύριε Κύρχο, ευχαριστούμε για τις φιλοφρονήσεις και τα σχόλιά σας για το τρίο των προεδριών και Ευχαριστώ γενικότερα του συναδέλφου για τα καλά τους λόγια. Για τη ριζοσπαστικοποίηση έχουν γίνει πολλά από πλευρά και του Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Υπάρχει η ειδική μονάδα στη Europol για το διαδίκτυο. Σημαίνει ήδη ε, επιτυχία η δράση της και χρησιμοποιούνται εμπειρίες ε, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τους συναδέλφους μας. Για τη ρισοσπαστικοποίηση συνειδητοποιεί το Συμβούλιο ότι σε αυτό το τομέα όλος ιδιαίτερος θα πρέπει να επιδιώξουμε την ανταλλαγή πληροφοριών για τα κηρύγματα μίσους, για τα μηνύματα μίσους, στις 2 ε, Φεβρουαρίου έχουμε την πλήρη προσέγγιση για τον ε, βίο εξτρεμισμό και ριζοσπαστικοποίηση, ε, μια διάσκεψη που θα συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Η κυρία Σατζεντίνη επίσης το ίδιο ρώτησε για τα κηρύγματα μίσους. Το συζητήσαμε στο Συμβουλίο και αποφασίσαμε πρώτον να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και δεύτερον να έχουμε διμερείς επαφές για συγκεκριμένα άτομα που κηρύσουν το μίσος. σε συνδυασμό φυσικά με την ε, ειδική μονάδα για το διαδίκτυο και την ε, αντιτρομοκρατία στη Europol. Ε, η κυρία Βίξτρομ μας έρωτησε για το κράτος δικαίου και ο κύριος Διγιούγκ έκανε παρεμφερή ερωτήματα καθώς και η κυρία Σαρκεντίνη. Ε, σε σχέση με την, ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο, το κράτος ε, δικαίου, τη νομοθεσία για τα ΜΜΕ και τις εξελίξεις στην Πολωνία, έχουμε να πούμε πως ε, οι θεμελιώδει αξίε ε, θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ ε, σε ολόκληρη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθούμε του Συνεκέ στις επαφέ που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Πολωνική Κυβέρνηση και το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Την επόμενη Τετάρτη στο Σώμα των Επιτρόπων θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και ίσω μάθουμε περισσότερα για τη θέση τη Επιτροπής. Επίση, ανάμεσα στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και την Πολωνική Κυβέρνηση γίνονται ιδιαίτερα σημαντικέ επαφέ στα πλαίσια τη Επιτροπή Βενετία στα τέλη Ιανουαρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια το θέμα της Πολωνίας και τονίζεται έτσι η σημασία ε, του θέματος αυτού. Ο Υπουργός εξωτερικών κουνής θα παρευρεθεί στη συζήτηση και με ρωτήσατε αν θα έρθω σε επαφή με τον Πολωνό ομότιμό μου. Φυσικά, ε, στα πλαίσια της ε, θα έρθω σε επαφή μαζί του για μια σειρά ζητημάτων αλλά και για ε, τυχόν ανησυχίες που έχουμε ε, σε σχέση με το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Κυρία Σίπελ, μου έκανε μια ερώτηση για το κυβερνοέγκλημα. Με ρώτησε αν έχουμε ε, ορισμό. Αν τον είχαμε, θα σας τον είχαμε κοινοποίησει. Ε, όλοι αντιλαμβάνονται με κάποιο τρόπο ε, το κυβερνοέγκλημα, αλλά όλα αυτά ε, είναι δεν αποτελούν ορισμό, διότι υπάρχουν επικαλύψεις με, άλλα, με είναι μεγάλη πρόκληση όντως αυτό. Επίσης ε, μας είπατε ε, για τη ληστεία, ναι ξέρουμε ποιος είναι ο εισαγγελέας ο οποίος θα διώξει ε, το αδίκημα. Όμως όταν γίνει το έγκλημα στη Γαλλία και ο εγκληματίας είναι στη Γερμανία και το θύμα ζει στην Ελλάδα, τότε έχουμε θέματα δικαιοδοσίες. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θέλουμε να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε τους επόμενους έξι μήνες. Επίσης, ε, ρωτήσατε για ε, την, ε, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το θέμα της χρηματοδότησης. Φυσικά έχουμε πλήρη επίγνωση το ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε ευρύτερα το ζήτημα διότι δεν θέλουμε να χρηματοδοτούνται καθόλου οι τρομοκρατικέ οργανώσει. Θέλουμε να διακοπεί η χρηματοδότηση. Κύριε Ντογιόνγκ, επιβεβαιώσατε και σα ευχαριστώ γι' αυτό πω και εσεί προτίθεστε να συνεργαστείτε μαζί μα ε, ώστε να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για την νομική συνδρομή. Προσβλέπω στις ε, επαφές που θα έχουμε μελλοντικά για αυτό το ζήτημα. Ε, κύριε Σαγετίνη, με ρώτησε για την Ουγγαρία και για την απόφαση ε, του δικαστηρίου. Τι έγινε. Ένας ε, Ολλανδός ε, δικαστής ανέβαλε την μεταφορά των κρατουμένων περιμένοντας την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε λοιπόν να εκδοθεί η απόφαση και μετά από αυτό θα αντλήσουμε τα δάγματα και θα βγάλουμε συμπεράσματα και θα λάβουμε υπόψη και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είναι εφαρμοστό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Κυρία Φεράρα. Ρωτήσατε για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών κατά πολέμηση τρομοκρατίας. Ε, από την περσινή μου εμπειρία στο Συμβούλιο θα έλεγα πως τα κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό είναι πεπισμένα για την σημασία που έχει η ανταλλαγή πληροφοριών. Στο άτυπο ε, Υπουργικό Συμβούλιο θα ε, συγκεκριμένα για τους εκπριστοκροτητές και τα πυροβόλα όπλα θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και στα πλαίσια των εθνικών στρατηγικών και Νομίζω ότι στο Συμβούλιο υπάρχει ομοφωνία σε σχέση με το ε, κέριο ρόλο που έχει ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση και τη οργανωμένη εγκληματικότητα αλλά και τη τρομοκρατία και φυσικά έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού. Θα δώσω, νομίζω, Πρόεδρε, α, μην ανησυχείτε, θα έχετε και άλλες ερωτήσεις, γιατί ακολουθεί και άλλος γύρος. Ο κύριος ε, Ντάικοφ ε, Ξέρω ότι είναι πολλές οι ερωτήσεις, μην ξεχνάτε όμως ότι για τη μετανάστευση θα σας απευθύνουν περισσότερες ερωτήσεις για τα θέματα μετανάστευσης στον επόμενο γύρο. Ίσως 5-6 λεπτά για να απαντήσετε στους συντονιστές θα έλεγα. Εντάξει λοιπόν, ε, δεν θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος να απαντήσω τις εύκολες ερωτήσεις και να πω άμετα πάνε τα 6 λεπτά». Ε, νομίζω ότι αρκετές ερωτήσεις ετέθησαν ε, από εσάς όσον αφορά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και τι έχουμε καταφέρει και τι δεν έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι καλό είναι να πούμε ότι αν δείτε αυτή τη στιγμή τα αριθμητικά στοιχεία, ε, αν δείτε τι έχουμε συμφωνήσει, η μετεγκατάσταση δεν είναι καν ε, δυνατή αυτή τη στιγμή. Μπορούμε απλώς να κάνουμε μεταφορά. Η μετεγκατάσταση σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει αρχικά υποδοχή, γίνεται η καταγραφή και εμείς αυτή τη στιγμή το χτίζουμε αυτό σιγά σιγά. Πρέπει να δημιουργηθούν όλα τα hot, stop, hot spots και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής ε, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε χτυλικά αποτυπώματα και να συμπεριληφθούν σε ένα σύστημα το οποίο από εκεί και πέρα θα είναι ένα σύστημα στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια ανάλυση των προσφύγων, ε, ε αναπερίπτωση και όχι βάσει του συνολικού αριθμού αιτήσεων ε, ασύλων, ε, αλλά να δούμε κατά πόσον ε, βρίσκονται στο πλαίσιο, στην κατηγορία του 75% είναι ε, ε, πιθανότητες ε, να λάβουν τη καθεστώς πρόσφυγα, αν έχουν οικογένεια σε κάποια χώρα, αν υπάρχει δηλαδή ένα λογικό χώρο στον οποίο θα μπορούσαμε να μετεγκαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, αυτό ε, σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, προσπαθούμε να δοκιμάσουμε το σύστημα μένα, αλλά και να το βελτιώσουμε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη Ολλανδική θέση, ξεκινήσαμε με δύο hot spots για την Ιταλία και για την Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε την πρώτη εβδομάδα να έχουμε άφηξη των πρώτων ανθρώπων και την πρώτη μετεγκατάσταση, αλλά δεν είναι η διαδικασία μετεγκατάσταση όπω την είχαμε προβλέψει αρχικώ. Αυτή δεν την έχουμε αρχικά. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να λειτουργούν αποτελεσματικά όλα τα hot spots ε, από, ε, ε, για να ξεκινήσουμε. Είναι μια διαδικασία όμως που είναι δυτή. δεν σημαίνει απαραίτητα όμως ότι όλοι βρίσκονται στην πρώτη χώρα άφηξης. Ε, υπάρχει ένα ανεπίσημο σύστημα μετεγκατάστασης. Ε, ε, κάποιοι φτάνουν σε μια χώρα και είτε όχι, καταγράφονται είτε όχι, φεύγουν και μετεγκαθίστανται μόνοι τους. Εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία καταγραφής τους. Επομένως, εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω απογοητευτεί περισσότερο από όλους για τους ρυθμούς, αλλά δεν ε, ε, λέω τόσα πολλά ε, όσα έλεγα πριν επισκεφθώ τα ελληνικά νησιά. Καταλαβαίνω αυτού που λένε ότι δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, πρέπει να ξεκινήσουμε και, ε, με και από το μηδέν. Σε κάποια νησιά χρειάστηκε να ξεκινήσουμε από το τίποτα. Δεν λέμε ότι ξεκινάμε από ένα σύστημα που λειτουργεί και απλώ πρέπει να κάνουμε κάποιε προσαρμογέ. Είναι πολύ εύκολο να το λέει κάποιο ε, απ' έξω όταν τα βλέπει τα πράγματα. Λέει γιατί παίρνουμε δαχτυλικά αποτυπώματα σε χαρτί και όχι σε ένα σύστημα υπολογιστή. Γιατί δεν υπάρχουν ε, ε, συστήματα υπολογιστή σε όλα τα νησιά. Υπάρχει ένα πλεόνισμα λοιπόν το οποίο δεν καταγράφεται ούτε με τον παραδοσιακό τρόπο ούτε σε σύστημα υπολογιστή και επομένως ε, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι έχουμε ξεκινήσει και γίνεται πολύ καλή δουλειά και έχουμε πετύχει ένα θαύμα. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία γιατί υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου που ε, θα έπρεπε να ε, εγκρίνουν την πρόταση νωρίτερα, ίσως έτσι να είχαμε και λίγο περισσότερο χρόνο και όσον αφορά τις ερωτήσεις που έγιναν ε, για το μέλλον της Σέγγεν και αυτές τις πολύ γνωστές ιδέες, δεν θα μπορούσα να τις αποκαλέσω προτάσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή να τις αποκαλούμε προτάσεις αυτές τις προτάσεις για τη μήνυ Σέγγεν. Ε, συζητήθηκαν σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και στις κάτω χώρες. Δεν είναι πρόταση, δεν είναι στόχος. Ο στόχος είναι η Σέγγεν. Η Σέγγεν είναι το καλύτερο που έχουμε. Δεν πρόκειται για σχέδιο Α, ούτε σχέδιο Β, ούτε σχέδιο Γ ούτε αμφισβητεί κάποιο τη Σέγγεν ε, λόγω τη έλλειψη πολιτική απόφαση από πλευρά κρατών μελών. Νομίζω ότι την άνοιξη του 2015 ε, υπήρχε ήδη ανάλυση ότι αν δεν καταλήξουμε σε κάποιε λύσει τι οποίε θα εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη ή τουλάχιστον όλα τα κράτη-μέλη τη Σέγγεν, κινδυνεύει η συνθήκη Σέγγεν. Είναι μια ανάλυση, δεν είναι επιθυμία, κάθε άλλο. Εμείς επιθυμούμε ακριβώς το αντίθετο δεν καταφέραμε εμείς τα κρατημένα να συμφωνήσουμε και επομένως η απειλή ε, είναι πλέον ε, κάτι το οποίο είναι πιο σοβαρό, δεν είναι ανέκδοτο. Πρέπει οι χώρες να συνεργαστούν, δεν μπορεί να αφήνουν η μία χώρα του, όλο τον κόσμο να περάσει για να αναλάβει μία χώρα την υποδοχή. Ε, και βλέπουμε ότι μπορεί να ξεκινήσει και ο πανέλεγχος στα σύνορα. Εάν χρειάζονται κάποιες χώρες ε, δικαιολογία θα μπορούσαν να το είχαν κάνει πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι δεν θέλουν οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, δεν το κάνουν γιατί τους αρέσει, αλλά γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Και όσον αφορά τη δυνατότητα να έχουμε ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκη, είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κάποιος ότι θα πρέπει να υπάρχει κατανομή βαρών από του 28. Θέλουμε να γίνεται κατανομή των ροών με καλύτερη συνεργασία στις χώρες της περιοχής. Ε, αυτές οι συνδυασμένε προσπάθειες είναι το πρώτο μας σχέδιο και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορε άλλε εναλλακτικέ λύσει. Ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία στα θέματα αυτά και μετά ε, είναι λογικό κάποιες χώρες να σκέφτονται ε, τι θα γίνει αν δεν λειτουργήσει αυτό. Ε, ξαναλέω, δεν είναι ούτε σχέδιο Α, ούτε σχέδιο Β, ούτε σχέδιο Γ. Δεν είναι μια πρόταση, είναι ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Δεν θα το προωθήσουμε αυτό γιατί προτιμούμε όλες τις άλλες λύσεις, αλλά εάν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε λύσεις, δεν μπορεί οι κυβερνήσεις απλώς να πούνε ότι α, δεν έχουμε ε, το σχέδιο Α, άρα δεν θα κάνουμε τίποτα. Ε, σίγουρα πρέπει να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση, αλλά δεν είναι λογικό να νομίζουμε ότι θα μείνουν αδρανή τα κράτη-μέλη. Πρέπει να έχετε μια ιδέα λοιπόν του σε τι πλαίσιο συζητήθηκε. Όχι προτάθηκε, αλλά συζητήθηκε. Ε, τουλάχιστον αυτό διέρευσε ότι συζητήσετε. Ο Πρόεδρος, θέλουμε να μάθουμε πολύ περισσότερο για το θέμα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Ε, και γνωρίζω από τον κατάλογο των ομιλητών μου ότι οι αρκετοί συνάδελφοι θα σας θέσουν ερωτήσεις για τη μετανάστευση και για τη Σέγγεν. Θα ήθελα λοιπόν να τους δώσω το λόγο και από εκεί και πέρα ε, μπορεί να πούν και κάποια συμπληρωματικά σε αυτά που είπατε. Θέλω λοιπόν να συνεχιστεί ο διάλογος, να μιλήσουν όλοι, θα μπορέσετε να μείνετε τουλάχιστον μέχρι τις 5 και ίσως ε, λίγο αργότερα ο κύριος Βαντεστήρ θα πρέπει να φύγει στις παρατέταρτο. Επομένως θα ήθελα να δώσω τους λόγους στους συναδέλφους και από εκεί και πέρα θα έχετε εσείς περισσότερο χρόνο για να συζητήσετε αυτά που λέτε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ομπόνη. Συνάδελφοι, ε, δύο λεπτά σας παρακαλώ για να βοηθήσετε και μενωμένα. Ευχαριστώ πολύ και θα μιλήσω πολωνικά. Κύριοι Υπουργοί, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρουσιάσεις σας των προτεραιοτήτων της Ελλανδικής Προεδρίας. Οι πτυχές αυτές προστασία συνόρων, χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία των συνόρων μας, ε, διαφύλαξη του Σέγγεν, νέες ε, αντιτρομοκρατικές οδηγίες, ανταλλαγή πληροφοριών έχουν κέρια σημασία και έχουμε νομίζω αφήσει να περάσουν εβδομάδες και μήνες κρίσιμοι. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία λοιπόν, συνεργασία που δεν υπάρχει. Και εδώ έχουμε ζητήματα και με το κράτος δικαίου ακούσει να και εγώ προερχομένως από την Πολωνία θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Υπουργό Στέρ για την πολύ ψύχρεμη ενημέρωση που μας έδωσε. Μας είπατε ότι θα ασχοληθείτε με τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τα ζητήματα και τα όσα συμβαίνουν στην Πολωνία. Πιστεύω ότι το κράτος δικαίου το θέμα του ε, συνταγματικού δικαστηρίου έχει υπονομευθεί ιδιαίτερος ε, χρειάζεται συζήτηση. Υπάρχουν συζητήσεις και στην Επιτροπή της Βενετίας έχουν άλλωστε παραβιαστεί και άλλοι κανόνες. Θέματα που έχουν να κάνουν με την ανεξαρτησία των δημοσίων υπαλλήλων, Και υπάρχουν και κριτήρια σχετικά με τα υψηλότερες θέσεις αξιωματοχών της δημόσιας διοίκησης που πρέπει να κοιτάξουμε μεγαλύτερη προσοχή. Υπάρχει και άλλο ζήτημα που προκύπτει, νομοθεσία σχετική με την αστυνόμευση, η οποία ανατρέπει τις ισορροπίες μεταξύ προστασίας ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχουν κριτήρια φερρυπίν των πιο σοβαρών αδικημάτων ε, και προβλέπεται η δυνατότητα διώξεων εις βάρος ε, πολιτών χωρίς ε, διάκριση βαρύτητας αδικημάτων. Με μεγάλη λύπη τα επισημαίνω όλα αυτά και πιστεύω ότι θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες και ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, αγαπητή συνάδελφοι, σας παρακαλώ μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά. Κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους υπουργούς από πλευράς κάτω χωρών για το πρόγραμμα το οποίο μας παρουσίασαν και να ευχαριστήσω ιδιαίτερος ε, τον ε, κύριο Φαντεστέρ για την ε, παρουσίαση που μας έκανε για την οδηγία για τους ανηλίκους, ε, στην οποία ήμουν εισηγήτρια και που θα ήθελα να πω ότι είναι αποτέλεσμα της συνεργασία με τους κοιόδη συζητητέ αλλά και της δέσμευσης της Λουξεμβουριανή Προεδρίας για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ήθελα να ενθαρρύνω και την Ολλανδική Προεδρία να προχωρήσει ε, ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία και για την οδηγία για την νομική συνδρομή του συναδέλφου Ντεγιόγκ ώστε να ολοκληρώσουμε τον οδικό χάρτη για τις ε, διαδικαστικές εγγύησεις. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν θα ήθελα να κάνω δύο πολύ σύντομε παρατηρήσεις. Η μία αφορά την τρομοκρατία. Όσον αφορά την τρομοκρατία, δεν άκουσα να συζητείτε πολύ. Ο Τη πρόληψη, που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη για τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω κατάλληλη μόρφωση, εκπαίδευση, στα σχολεία, μέσω τη πρόληψη και στα σοφρονιστικά καταστήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά την τρομοκρατία υπάρχει και ένα, μια άλλη πτυχή που είναι οι ε, δραστηριότητες ε, της υπόγειας εγκληματικότητας η οποία χρηματοδοτεί ε, δυστυχώς την τρομοκρατία αλλά και με συγκεκριμένε πράξει, όπω για παράδειγμα την παράνομη διακίνηση όπλων. Όσον αφορά όμως το οργανωμένο έγκλημα εν γέννη, πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων, ε, διότι ε, το οργανωμένο έγκλημα είναι αυτό το οποίο ε, χρηματοδοτεί. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα το οποίο υποστηρίζει την τρομοκρατία και υποστηρίζει και την ε, μετανάστευση, τη μεταφορά τρομοκρατών. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν ακόμα και θα ήθελα να σας ε, κάνω αυτή την παρατήρηση και να ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And... Σας ευχαριστώ. Κύριε Νιτφέλτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Φάντερστερ, κύριε Ντάικοφ, χαίρομαι που μπορώ να σας συναντήσω εδώ και βέβαια προβλέπω στη συνεργασία στο επόμενο εξάμεινο. Λίγο χρόνο έχω. Μια ερώτηση λοιπόν που αφορά τους πρόσφυγες καταρχάς. Δεν σας κρυβώ ότι ακούω πολύ να γίνεται λόγος για το θέμα των προσφύγων και το πόσο δύσκολη είναι η επίλυσή του. Δύσκολο θέμα, ναι αλλά δεν είναι και ανεπίλητο. Έχουμε χάσει χρόνο γιατί δεν θέλησαν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν την ευθύνη της επίλυσης και ελπίζω στο δικό σας εξάμεινο να εκφραστεί πολιτική βούληση. Δεν χρειάζεται να συστήσουμε λεπτομερώς ε, τις λύσεις ή τις λεπτομέρειες των λύσεων. Θέλουμε όμως να ξέρουμε ότι έχετε διάθεση να εξασφαλίσετε ομόφωνη στάση και δράση των 27 κρατών μελών για την Πολωνία και την Ουγγαρία. Όταν έρχεται το θέμα αυτό, πολύ συχνά λέγεται ότι πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις, monitor, ε, κοιτάμε την, ε, ε, να περιμένουμε την έκβαση των μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με χαρά ακούω ότι ενδιαφέρεστε για το θέμα της Πολωνίας. Το Συμβούλιο όμως έχει κάνει δική του αξιολόγηση κατάστασης. Δεν θα πρέπει να μην περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να του υποδείξει τι πρέπει να ε, αποφασίσει. Θέλω λοιπόν τις δικές σας σκέψεις και ιδέες από το Συμβούλιο. Για το κράτος δικαίου και τον διάλογο των σχετικό με το κράτος δικαίου, ιδιαίτερος χαίρο για τα πρώτα βήματα που πραγματοποιήθηκαν, αλλά ε, είναι κάπως ε, ελαφριά αντιμετώπιση της σοβαρότητας του κράτους δικαίου ή διεξαγωγή συναντήσεων και συνεδριάσεων μια φορά το εξάμεινο χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή και να μιλήσουμε πολύ πιο απερίφραστα προς εκείνα τα κράτη τα οποία φαίνεται να αδιαφορούν για το κράτος δικαίου και όπως υπόθηκε μόλις τώρα όταν ε, υπάρχει παρακολούθηση σε σχέση με το θέμα του ε, εντάλματος σύλληψης και την έκδοση και βλέπουμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης και η ε, έκδοση Πρέπει αυτά να, τα, να σας απασχολήσουν. Ο διάλογος για το κράτος δικαίου πρέπει να ενισχυθεί από την Ολλανδική Προεδρία. Και επίσης μια τελευταία ερώτηση. Τι θα κάνετε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η οδηγία κατά των διακρίσεων, που επί 10 χρόνια τώρα βρίσκεται σε τέλμα σχετικά με την αναγνώριση καθεστώτος ιδιοκτησίας και ε, των σχετικών με, τις, ε, ε, με τα σύμφωνα συμβίωση που παρεμποδίζουν συγκεκριμένα η Πολωνία και η Ουγγαρία. Τι θα κάνετε γι' αυτό, η κυρία Κέλλερ παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει κυρία Κέλλερ, για την μετεγκατάσταση. Εντάξει, η πρώτη φορά το δοκιμάζουμε, ναι, είναι δύσκολο, ναι, χρειαζόμαστε χρόνο, όμως αυτό δεν εξηγεί γιατί ε, ε, η Ολλανδία 100 θέσεις έχει μόνο προτείνει. Δεν εξηγεί γιατί ε, κάποια άλλα κράτη-μέλη ούτε μία θέση δεν έχουν προτείνει. Μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα από τους περασμένους μήνες. Πρώτον, ε, περιμένουν υπερβολικά πολλοί πρόσφυγες. Δύο μήνες ε, είναι πάρα πολύ. Κάπου πρέπει, να φτάσουν στον προορισμό τους ε, οι πρόσφυγες και κάπου πρέπει να μένουν για αυτούς τους δύο μήνες. Και αυτά τα κέντρα δεν κάνουν για δύο μήνες. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, όμως θα πρέπει να είναι ευέλικτα τα κράτη-μέλη. Κύριε Ντάικοφ, η Ολλανδική Προεδρία θα μπορέσει, θα θελήσει να προωθήσει αυτά τα ζητήματα. Δεύτερον, μιλήσατε για το για τους πρόσφυγες, για τον έλεγχο κατά την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους διακινητές, ε, για την ε, τραγική μοίρα των προσφύγων. Ε, ναι, εάν δεν έχουμε νόμιο εδώ διέλευση των συνόρων, χερσαίων συνόρων, πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να βρούμε λύση. Έτσι θα σώσουμε και πάρα πολλέ ζωέ. Ε, η Ολλανδική Προεδρία θα αναλάβει πρωτοβουλίε προ αυτή την κατεύθυνση για να καταστήσει ε, δυνατή την νόμιμη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφύγουμε τις ε, εκατοντάδες χιλιάδε προσφύγων από την Τουρκία παραδείγματο χάρη. Ευχαριστούμε κύριο Κύρκο. Thank you, Chair. Um, το πολύ ενδιαφέρον κείμενο της Ολλανδικής Προεδρίας βλέπουμε τις τρεις προτεραιότητες, δηλαδή την υποδοχή προσφύγων που σχετίζεται με τα hot spots, την προστασία των εξωτερικών συνόρων που σχετίζεται με τις επιστροφές και το διαμοιρασμό των βαρών που σχετίζεται με τη μετεγκατάσταση. Λαμβάνουμε υπόψη βεβαίω ότι τα hot spots δεν είναι στη θέση του παρόλο που θα έπρεπε να είναι από τον Οκτώβριο πως η πολιτική των επιστροφών δεν υπάρχει. Πριν από λίγες εβδομάδες ένα αεροπλάνο από την Ελλάδα πήγε στο Πακιστάν και γύρισε με τους μισούς Πακιστανούς υπηκόους μέσα γιατί η κυβέρνηση δεν τους δεχόταν πίσω και απλώς ο μηχανισμός κατάσταση δεν λειτουργεί. Ξέρουμε λοιπόν πως στο εξάμεινο που έρχεται θα περάσουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τα θαλάσσια σύνορά μας. Σε έξι μήνες θα έρθετε να δούμε τα αποτελέσματα της Ολλανδικής Προεδρίας. Και μια ιδανική περίπτωση θα ήταν το 100% των ανθρώπων που φτάνουν στις ακτές μας να είχαν φιλοξενηθεί με συνθήκες αξιοπρέπειας, να είχαν όσοι δικαιούνται ε, μετακινηθεί σε άλλες χώρες για να διερευνηθεί η άδειά του περί ασύλου και όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να μετακινηθούν να επιστραφούν στι χώρε του. Αυτό ήταν το ιδανικό. Αν, μας, αν κάποιο μα έλεγε ότι ναι, αυτό είναι το ιδανικό, αλλά εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα καταλαβαίνουμε πω πραγματικά δεν υπάρχει ένα σχέδιο, δεν υπάρχει κάποια γνώση τη κατάσταση, υπάρχει απλώ μια καλή θέληση. Εμεί θέλουμε από εσά, κύριε Ντάικοφ, όχι να μοιραστείτε τον τρόμο σα μπροστά στο πρόβλημα, τον ίδιο τρόμο έχουμε κι εμεί, γιατί ξέρουμε πω η Ευρώπη δεν θα αντέξει άλλο ένα καλοκαίρι σαν αυτό που πέρασε. Αυτό που θέλουμε είναι με αριθμού να μα δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα πότε προβλέπονται να ισχύσουν τα hotspots. Όχι όλα, γιατί το hotspot της νήσου ΚΟ δεν θα υπάρξει, όπως έχει πει και ο Υπουργό. Πότε θα υπάρξει η μετεγκατάσταση, πότε θα ξεκινήσουν οι πολιτική των επιστροφών. Αριθμούς θέλουμε, τις δικές σας δεσμεύσεις πάνω στην προεργασία που έχετε κάνει για να αναλάβετε την Προεδρία. Γιατί δεν είναι μόνο ένα όμορφο κείμενο να λαμβάνουμε, είναι αυτό το κείμενο και ελπίζουμε να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Kiangi, please. Η κυρία Κέγκη. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάω από το θέμα το οποίο επενθύμησε και η συνάδελφος ε, Ρομπέρτα Μέτσολα. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί η έκθεση στρατηγικής πρωτοβουλίας η οποία θα αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης ε, ζητώντας ε, να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση. Σε αυτή την ε, έκθεση πρωτοβουλία θα περιλαμβάνονται πολλά από τα σημεία τα οποία μα παρουσιάσατε και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θα ήθελα να κάνω κάποιε ερωτήσει. Καταρχά, αυτή είναι μια ελπίδα που εκφράζω. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά στη διάρκεια της Προεδρίας σας για το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί την επίσημη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μετανάστευση. Δεύτερον, αναφερθήκατε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κρατημέλη για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ροών. Πώς σκοπεύετε να βοηθήσετε εσείς τα κρατημέλη; μελη αυτά. Και επίσης πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το θέμα της ε, Επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα, το οποίο ε, αναφέρεται όλο και πιο συχνά και γίνεται όλο και πιο συχνά. Ε, το ανέφερε και κάποια άλλη συνάδελφος. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει συζήτηση για αυτή τη μίνι Σέγγεν. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω εάν συζητάτε περισσότερο από ό,τι γνωρίζουμε γι' αυτό. Και ένα τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να ε, σας θέσω. Δεν άκουσα τίποτα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, ε, της Ισλαμοφοβίας και του ρατσισμού. Ε, ηθελημένα δεν έχετε αναφέρει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στίβενς. voorzitter en collega's en Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να σας κάνω μια ερώτηση για την μετανάστευση. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε για αυτό το ζήτημα, θεωρείτε πως οι πρόσφυγες που πηγαίνουν προστασίας στην Τουρκία θα ε, επαναπροωθηθούν επίσης ή όσοι έρθουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δικαιούνται προστασία. Επίσης, σε συζήτηση με τον κανονισμό του Δουβλίνου προβλέπετε πως η πρώτη χώρα είναι υπεύθυνη και για την ε, υποδοχή. Αλλά φυσικά βλέποντας την κατάσταση στην Ιταλία και στην Ελλάδα, συνειδητοποιούμε ότι είναι αφόρητη η κατάσταση. Λοιπόν, προβλέπεται κατανομή και βάση ποιας κλίδας ε, αυτής που έχει αποφασιστεί ή μήπως έχετε νέες ιδέες να καταθέσετε. Φυσικά δεν είναι ε, λύση η απόρριψη του Δουβλίνου, αλλά τι αντιπροτείνεται. Ευχαριστούμε κυρία Νταλή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ολλανδική Προεδρία για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων. Δεν θέλω να επανέλθω στο μηχανισμό κατάστασης, διότι ακούσαμε ήδη πολλά ερωτήματα για αυτό το ζήτημα όμως αφήσατε αναπάντητα πολλά ερωτήματα. Τουλάχιστον εγώ δεν ικανοποιήθηκα από τις ερωτήσεις. Είμαι από τη Μάλτα. Διάβασα το πρόγραμμα των τριών προεδριών και χάρηκα διότι τονίζατε τη σημασία της ευθύνης των κρατών μελών και της αλληλεγγύης. Είναι αργές οι εξελίξεις, ομολογουμένως. Ταυτόχρονα όμως ε, είναι και περιορισμένα τα μέσα. Όμως δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αυτό ως ε, πρόσχημα για να μην κάνουμε τίποτα. Για τους ε, σοσιαλιστές είμαι εισηγήτρια για το θέμα της μόνιμης επανεγκατάστασης και θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για αλληλεγγύη μακροπρόθεσμα εάν ακόμη και για τα προσωρινά μέτρα δεν μπορούμε να, δείξουμε, να επιδείξουμε την απαιτούμενη αλληλεγγύη. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω για την Ολλανδική Προεδρία και το Τρίτο των Προεδριών ναι, ποιες δράσεις συγκεκριμένα θα αναλάβετε Κύριε Βαντεστέρ, μιλήσατε και για την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων για την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας. Αυτό έχει καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση των δικτύων στην Ευρώπη και εσείς προτείνετε μια ολιστική προσέγγιση για την οργανωμένη εγκληματικότητα και τους διακινητές. Πώς θα ακριβώς, τι θα κάνετε στην πράξη για να υπάρξει και ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, ασφάλεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νίτερμελ. Ε, μας ε, παρουσιάσατε τις προτεραιότητες ε, της Προεδρίας. Καλωσορίζουμε τις ιδέες σας και την πρότασή σας για συνεργασία. Το κράτος δικαίου είναι βασικό πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθεροτυπία, συνταγματικές ελευθερίες δεν τίποτα για κάποιες χώρες. Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η Ουγγαρία και η Πολωνία, μη φιλελεύθερες, ανελεύθερες δημοκρατίες. Ε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας αποτελεσματικότερος μηχανισμός παρακολούθησης ε, διότι υπάρχουν διατάξεις όμως ε, δεν, υπά, δεν προτείνεται καμία αλλαγή σε αυτές τις χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα κράτους δικαίου. Λοιπόν, σας ρωτώ τι ακριβώς θα κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας όπου καταπατώνται βασικές ελευθερίες. Περιμένουμε πολλά περισσότερα από το Συμβούλιο. Τι σχεδιάζετε συγκεκριμένα να κάνετε για να διαφυλάξετε το κράτος δικαίου ε, σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Βίνμπεργκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Το 2016 θα είναι ιστορικό έτος ε, σε σχέση με την αντίληψη του κόσμου και σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε και τις ευθύνες που καλούμαστε να υπομειστούμε. Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ε, αυτή τη στιγμή όποια μέσα έχει για να αντιμετωπίσει τα, τους χαμηλότερους σχετικά ρυθμούς προσφύγων διότι είναι η χειμερινή ε, περίοδος και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ κακές επιδόσεις από χώρες όπως και η Ολλανδία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού κύματος. Τι μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν τις επόμενους έξι μήνες για το μηχανισμό κατανομής. Πώς, θα Πώς τελικά θα εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτών που έχουμε συμφωνήσει. Τι, θα υπάρχουν πρόστιμα, θα υπάρχουν κυρώσεις, το έχετε σκεφτεί καθόλου για τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν τα μέτρα. Ε, τι θα κάνουμε τώρα με αυτούς που έχουν πάει στη Συρία και επιστρέφουν τώρα, ε, θα, ε, πέρα από ε, τον όλο διάλογο για τη ριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη. Συγκεκριμένα θα υπάρξουν αποτρεπτικές κυρώσεις ε, κατά αυτών των ανθρώπων. Παραδείγματο χάρη ε, έρχονται αυτοί και κατατρομοκρατούν συμπολίτε μας. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι. Ε, τώρα, το κάτι άλλο, η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Υπάρχουν προτάσεις για τροποποίηση του κανονισμού εμάς ε, θα μας επηρεώσει πάρα πολύ αυτή η τροποποίηση. Θα παραβιάσει τα δικά μας δικαιώματα στη Σουηδία. Πώς το βλέπετε εσείς, κυρία Μπιόρκ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι δίκιο έχετε όταν λέτε ότι υπάρχει κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλά τα λέτε, διότι ε, αποτύχαμε σε σχέση με αυτά που περιμένουν οι πρόσφυγες, αυτά που περιμένουν ε, αυτοί που θέλουν να ε, είναι πιο υπεύθυνοι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα έχουμε καταφέρει και όπως είπε και ο συνάδελφος, αλλά και στο, στη Δουνκέρκη, αλλά και στο Καλέ, βλέπουμε πλήρη αποτυχία. Δεν είναι τρόπος μεταχείρισης ανθρώπων αυτός και δεν δίνει απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ήρθε η στιγμή να δείξουμε πως δεν ε, θα αφήσουμε τους ρατσιστές να αποφασίζουν. Δεν θέλουμε περισσότερο χειρό Ευρώπη. Δεν είναι αυτό το μέλλον. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες ε, για να ενισχυθούν η διαφύλαξη των ε, σύνορων και τι σημασία έχουν αν δεν μπορούμε να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε τις εγκαταστάσεις, υποδοχή και μεταχείριση των φακέλων των εκατομμυρίων που ε, χρήζουν προστασία και δικαιούνται το καθεστώ. Έχουμε δυνατότητα βάσει των συνθήκων να προχωρήσουμε περισσότερο με ένα μικρό συνασπισμό χωρών που προτίθεται να κάνουν τα απαιτούμενα αυτή τη στιγμή. Επίσης, η ύπατη αρμοστία μπορεί να βοηθήσει, το ΙΕ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που θέλουν να προχωρήσουν, ε, να προχωρήσουν, να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει και ε, σε σχέση με αυτά που είπατε για την Ουγγαρία και την Πολωνία, κύριε Νιντερμάγερ, θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ. Είναι βασικότατο ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Αλλιώς θα υπονομεύεται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου από κάποιους και ενισχύουμε έτσι τις δυνάμεις της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Υπουργός Βαντεστέρ πρέπει να φύγει στις παρατέταρτο. Οπότε ε, θα δώσω το λόγο. Ε, κύριε Ντάικοφ, εσείς θα παραμείνετε λίγο παραπάνω. Άλλοι δύο και θα κλείσω τον κατάλογο, αν μου επιτρέπετε. Κυρία Ρεβού, Νταλόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και για άλλη μια φορά θα διατυπώσω και εγώ ερώτηση σχετική με το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Έγινε πολλής λόγος για την Πολωνία, αλλά και για την Ουγγαρία. Και ο κύριος Νίτερ Μιούλερ ε, της ανέφερε. Ε, θέλω να επανέλθω λοιπόν σε αυτή την κατάσταση με τις ε, ταχύρυθμες διαδικασίες που αφορούν τους πρόσφυγες, που τους απευθύνονται κατηγορίες Παράνομη ζέβαση συνόρων. Ε, Σλοβενία επίσης όπου ο Πρωθυπουργό λέει ότι πρέπει να παρακολουθούνται οι μουσουλμάνοι συλλήβδινο πιθανή απειλή για την τρομοκρατία. Τη Δανία σε σχέση με τη χρηματοδότηση της ε, υποδοχής των προσφύγων που θέτει όρια στι 3.000 κορώνες. Τη Σουηδία σε σχέση με τους ελέγχου ε, στα σύνορά τη με τη Δανία Πολλά είναι τα παραδείγματα και πολλά είναι τα ρήγματα σε σχέση με το κράτος δικαίου που διαπιστώνουμε. Ακούω λοιπόν ότι είπατε πώς θέλετε το Μάιο να κάνετε μια έκτακτη σύνοδο για το θέμα αυτό, μια Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν όμως των συζητήσεων και των προτάσεων χρειάζονται πράξεις συγκεκριμένα. Τι σκοπεύετε να πράξετε. Ξέρω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε το επίπεδο των ομιλιών και των τοποθετήσεων πρέπει να υπενθυμίσουμε τις αξίες μας και να τις υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ ο κύριος ε, Τζάζικ εν τέλει. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω μια ερώτηση που αφορά το κατά πόσον έχετε αναλογίσει τη δυνατότητα αξιοποίηση εφαρμογή τη οδηγίας προσωριν, περί προσωρινή προστασίας, τη οδηγία του 2001 σε σχέση με την κρίση των προσφύγων. Ε, πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο πιστεύω έχει σχεδιαστεί ακριβώς για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, τουλάχιστον σε σχέση με το Συριακό. Ο Πρόεδρος ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ συνεπείς στο χρόνο τους. Παρακαλώ τον Υπουργό Φαντεστόρ να κάνει σύντομες ε, τοποθετήσεις ε, σε ερωτήσεις που αφορούν κυρίως το κράτος δικαίου πριν αποχωρήσει. Πρόεδρε ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Κινίτση καταρχάς για τις παρατηρήσεις της που αφορούν ε, την τρομοκρατία. Είναι ύψης της σημασίας ε, για το Συμβούλιο το θέμα αυτό. Το έχουμε σε πρώτη γραμμή στο πρόγραμμά μας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών στα τέλη Ιανουαρίου. Θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν προκειμένου να υλοποιηθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στα τέλη του προηγούμενου έτους και θα διεξαχθούν ακόμη δύο σύνοδοι υψηλού επίπεδου για την εγκαταπολέμηση της ρουσπαστικοποίησης. Η πρώτη, και εδώ συνυπογράφω τις ε, θέσεις της κυρίας Κινίτσι και η δεύτερη σύνοδος αφορά την ε, ε, μετακίνηση, τα ταξίδια σε χώρες για σε άλλες χώρες για διαπράξη τρομοκρατικών επιθέσεων και η κυρία Κέντζε αναφέρθηκε σε θέματα κράτους δικαίου, ε, η κυρία Νετφέλτ αναφέρθηκε στις, ε, στα σύμφωνα συμβίωσης. Στις 4-5 Δεκεμβρίου στη συνεδρίαση του προηγούμενου έτους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε συμφωνία σχέση με σε, μια συμφωνία για ένα συμβαστικό κείμενο και ε, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι προτάσεις. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις διατάξει συνθήκες, αν θέλουν μπορούν να προχωρήσουν σε ενισχυμένη συνεργασία. Πρέπει να πω ότι όλο και περισσότερα είναι τα κράτη τα οποία έχουν, αποδεχθεί, έχουν αποστείλει τα αιτήματα τα σχετικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα αναμένεται πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κίνηση μια διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία. Και αν συμβεί αυτό, με την συνένεση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναλάβει δράση το Συμβούλιο. Κύριε Νετφέλτ, πρόκειται για ένα θέμα ύψης της προτεραιότητας προτεραιότητας για τις κατοχώρες. Κυρία Κέντζη, αναφέρθηκε στην ε, καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, της ξενοφοβίας. Ε, έχουμε προβλέψει να κάνουμε μια σύνοδο σχετικά με την ε, ομάδα εργασίας που ασχολείται με την καταγραφή και δίωξη των εγκλημάτων μίσους. Θέλουμε πάνω, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με την καλύτερη καταγραφή τέτοιων αδικημάτων και να βρούμε μοντέλα πρότυπα για τη λειτουργία της, ε, των δικαιοδοτικών οργάνων. Θα πρέπει να βρούμε μέσα ε, που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών. Κυρία Νετφέλτ αναφέρθηκε στην οδηγία κατά των διακρίσεων ο συνάδελφος θα αναφερθεί στο θέμα αυτό φαντάζομαι. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα όπως αντιλαμβάνεστε. Κυρία Ανταλή αναφέρθηκε στη λαθροδιακίνηση, στην διακίνηση ανθρώπων. Ε, υπάρχει διάσκεψη που βλέπετε στο Άμστερνταμ 18-19 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της οποίας ε, θα παρουσιαστούν και ιδέες πολυτομεακής συνεργασίας και κυρίως σχέση με την εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού από αυτά τα δίκτυα και βέβαια το λαθρεμπόριο εις βάρος ανθρώπων, τη λαθροδιακίνηση κράτος δικαίου και όλες οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν κύριε Πρόεδρε από τους ε, συναδέλφους βουλευτές δείχνουν πόσο μεγάλες ανησυχίες εκφράζονται και ε, απασχολούν το Κοινοβούλιο και το κράτος δικαίου. Βεβαίως, όπως είπα, το Συμβούλιο έχει ε, αντίληψη του το κράτος δικαίου αποτελεί υπεργονιαίο λίθο θα συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επιβεβαιώνοντας ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία και θέλουμε οι θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Το Μάιο θα ασχοληθούμε και με το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο. Το κλείσμα των συνόρων. Το Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, θέλει να ενισχύσει περισσότερο τι εκθετικέ σχέσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπουμε σε μια συνεργασία μέσα ευέλικτη σε, συνθήκε σε συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνη και σεβασμού. Και προσβλέπουμε εργασία αυτή. Ο πρόεδρο ήδη ανέφερα στου αδέλφου ότι πρέπει να πάτε στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, πολύ μικρότερη από τη δική μα, θα το γνωρίζετε ασφαλώ. Αλλά γνωρίζετε τι προτεραιότητές μα. έχετε τώρα μια ιδέα και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σχέση μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι απαντήσει που δώσατε σε όλε αυτέ τι ερωτήσει. Ε, αποχωρείτε εσείς και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ντάικοφ. Έχετε άφθονο χρόνο πλέον να απαντήσετε τις ερωτήσεις για τη μετανάστευση ε, που μας έχουν περισσέψει. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ ε, με την ησυχία σας τώρα και μπορείτε να επεκταθείτε στις ερωτήσεις που αφορούν και τη Σέγγεν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να τα εξισορροπήσω λίγο, να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις ε, μέσα στο δεκάλεπτο που έχουμε στη διάθεσή μας, να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Νομίζω ότι κάποιες ερωτήσεις ε, αφορούσαν ε, τι βάρος μπορούμε να αναλάβουμε. Να το θέσω ως εξής. Εγώ άκουσα δύο είδη ερωτήσεων ερωτήσεις που ετέθηκαν ε, ε, από τα κράτη-μέλη που έλεγαν ότι πρέπει να εμείς να κάνουμε το α και θα πρέπει να πείστε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν και κάποιοι άλλοι ρώτησαν πώς μπορεί να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για το οτιδήποτε. Ε, πράγματι, για μας είναι σαφές ότι δεν θέλουν το ίδιο πράγμα όλα τα κρατημέλη. Και επίσης, ως ε, Προεδρία του Συμβουλίου, εμείς ε, στόχο έχουμε να ε, κάνουμε προτάσεις τις οποίες θα μπορούσατε να καταλήξετε σε συμφωνία. Ε, καταλαβαίνω αυτό που λένε αρκετοί ότι είναι σπατάλη χρόνου να συντάσσονται ωραίες προτάσεις όταν ξέρουμε ότι δεν θα τις στηρίξει για παράδειγμα η Γαλλία για να περάσουν ή κράτη-μέλη που δεν θέλουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φυσικά είναι αρμόδια να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει ε, τήρηση των νόμων. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, νόμους και διαδικασίες και να ψηφίζουμε και μετά να έρχεται μια χώρα και να μας λέει δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν θα τα τηρήσω γιατί εφόσον αρχίσουμε και δεχόμαστε μια τέτοια λογική θα τορπιλήσει και όλες τις υπόλοιπε συμφωνίε που έχουμε κάνει. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να καταλήξουμε σε προτάσεις οι οποίες ε, θα λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις ανησυχίες. Διότι κάποιοι ρώτησαν και ε, αν, ε, πώς μπορούν να συμφωνήσουν οι χώρες για οποιοδήποτε νέο μηχανισμό μετεγκατάστασης. Ο πρώτος ήταν μία φορά σε περιορισμένο αριθμό και ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθεί συνένεση επ' αυτού πέρασε τελικά με ειδική πλειοψηφία και τώρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταφέρουμε τις χώρες να δεχτούν ε, προτάσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να εξετάζουμε ε, τους αριθμούς προσφύγων ε, και μεταναστών ε, μεταξύ των κρατών μελών και δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ρωτάμε τις χώρες αν μπορείτε να προτείνετε κάτι, αν έχετε κάποια ιδέα του τι σημαίνει να πάρουμε επιπλέον ανθρώπους, επιπλέον ανθρώπους που σκοπεύουν να έρθουν στην Ευρώπη, είναι τελείως διαφορετικό αυτό από το να προσπαθεί ε, να κάποιος να ξέρει ότι δεν είναι περιορισμένος ο αριθμός, ότι υπάρχουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, που όχι μόνο επιστρέφουν ανθρώπους που δέχονται ανθρώπους που ε, ε, εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν θα επιτρέπουν και σε ανθρώπους να φύγουν αν δεν έχουν φύγει με νόμιμα μέσα. Που σημαίνει βέβαια ότι δεν θα έχουμε μηδενική εισρωή στην Ευρώπη. Ε, χρειάζεται πολλή δουλειά, πρέπει να αναλάβουν ευθύνε και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου. εκτό της γεωγραφική μα επικράτειας σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερε ευθύνε στην ευρύτερη περιφέρεια όχι να λέμε ότι εντάξει τους έχουμε εκεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να τους προσφέρετε και κάτι, ε, ένα καταφύγιο, μια υποδοχή εκεί. Και πρέπει επίσης να έχουμε και ελέγχου στα σύνορα που θα επιτρέπουν ε, ώστε να έχουμε ε, πολύ μικρή ροή και με την κατάσταση να είναι απλώς ένας από τους ε, μία από τις νόμιμες μάλλον οδούς συγγνώμη, που μπορούμε να έχουμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό μας καθήκον, θα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να αντιληφθούμε όλες αυτές τις ροές ε, ε ανθρώπων και πώς μπορεί η κοινωνία μας να αντιληφθεί λίγο καλύτερα ε, τι βάρος της αναλογεί. Αν μπορέσουμε όλα αυτά να τα συμπεριλάβουμε σε μια σωστή συζήτηση, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε ευρύτερη συμφωνία και να μην έχουμε απλώς λίγες χώρες, και να πω επίσης ότι δεν είναι στόχος μας να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ λίγων κρατών μελών. Αυτό είναι αυτό που γίνεται τώρα, αν τα δείτε ειλικρινά τα πράγματα. Αν δείτε το μεγαλύτερο μερίδιο ε, προσφύγων, το έχουν αναλάβει πολύ μικρός αριθμός χωρών και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης ε, ε, και το εξή. Εάν χρησιμοποιείτε λανθασμένα επιχειρήματα και λανθασμένη ρητορία για μεγάλο διάστημα και παραπληροφορείτε του πολίτε σα και δεν πληρείτε τι ανθρωπιστικέ σα υποχρεώσει, ε, τελικά αυτό που θα γίνει είναι ότι θα πούνε ότι θα σας αφήσουμε εκτός συζήτηση ε, και ε, ε, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε. Αυτό δεν είναι σαν να προμεδετούμε αυτή τη συμπεριφορά και δεν νομίζω ότι θα πάμε προς αυτή την κατάσταση. Δεν είναι απλά τα πράγματα αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ στενό αλλά και το μόνο βιώσιμο περιθώριο για να έχουμε συμφωνίες. Κάποιος ρώτησε αν υπάρχει συμφωνία με τρίτες χώρες και παραδείγματο χάρη την Τουρκία. Το σκεπτικό δεν μπορεί να είναι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι, να υπάρχει διαδικασία τη μετεγκατάσταση, αλλά αν υπάρχει μια παράνομη οδό ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ρυθμίσουμε τα πράγματα ώστε να μην ε, έρχονται απεριόριστο αριθμό ανθρώπων ε, παράνόμω στην Ευρωπαϊκή Επιτεκράτεια. Το αυτό ισχύει και με τη λογική κάποιου που ρώτησε ότι αν συμφωνούμε ότι η χώρα υποδοχής δεν μπορεί να αναλάβει όλο το βάρος. Θα πρέπει ε, να έχουμε μετεγκατάσταση μόνο στην Ευρώπη. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό θα αποφέρει καρπούς. Ε. δεν μπορούμε να έχουμε ένα νέο σύστημα το οποίο ε, να μπορεί να βασίζεται απλώς σε μια πλειοψηφία, έστω και ειδική πλειοψηφία ή σε συνένεση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη με, λοιπόν και τις ανησυχίες που υπάρχουν χωρίς να θεωρούμε ως συμπέρασμα ότι επειδή υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες όλες οι υπόλοιπες χώρες δεν ε, συμμετέχουν και δεν χρειάζεται να αναλάβουν κανένα μερίδιο ευθύνης. Ε, το θέμα είναι πού θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ο κύριος Κυρκός ε, μας ρώτησε και μας είπε να μην γράφουμε απλώς μακροσκελή κείμενα, αλλά να έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όσον ε, αφορά τα hot spots, δεν είναι η έλλειψη χρονοδιαγραμμάτων το πρόβλημα, είναι ότι δεν ε, καταφέρει κανείς να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα. Και δεν αφορά μόνο απόφαση του Συμβουλίου. Αν θέλει κάποιος να την εφαρμόσει στην πράξη, ε, διαπιστώσαμε ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία δεν είχαμε προβλέψει εμεί ω Υπουργοί και αυτοί οι οποίοι κατάρτισαν τα χρονοδιαγράμματα, αλλά αφορά και τη διάθεση των κρατών να τους βοηθήσουμε και να δεχτούν να έρθουν και άλλοι να συμμετέχουν και να βοηθήσουν. Αυτό απαιτεί χρόνο. Είναι εύκολο να πούν οι κυβερνήσει ότι θα κάνουμε αυτό και αυτό, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάπως και την κατάσταση επιτόπου και τους ανθρώπους που ζουν εκεί, να τους εξηγήσουμε τι θα συμβεί ε, στην περίπτωση, για παράδειγμα, των ελληνικών hot spots ε, στα νησιά, να μπορέσουμε να έχουμε συνεργασία εκεί. Εμείς ως Προεδρία και ως χώρα μέλος είμαστε πλήρως διατεθειμένοι να βοηθήσουμε και την Ελλάδα και την Ιταλία με την εγκατάσταση αυτών των hot spots, αλλά δυστυχώς χρειάζεται χρόνο να διαπιστώσουμε και τι βοήθεια χρειάζεται, πότε ε, προσφέρεται, αν θα γίνει αποδεκτή επιτόπου. Ε, όταν πήγα, ε, συνάντησα συμπολίτε μου που ήταν εκεί αρκετούς μήνες και μου είπαν τι ακριβώς έχει γίνει, τι, πώς έχουν αλλάξει τα πρόβληματα τους τελευταίους μήνες, αλλά κανένας δεν ήταν επανευτυχής ότι τα έχουμε καταφέρει. Ε, είχαμε κάποια χρονογραμμάτα, είχαμε προθεσμίε, είχαμε ημερομηνίε οι οποίε είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουν το δικαίωμα να το κάνουν και να λένε ότι την τάδε μέρα θα, θα υπάρχει hot spot. Αλλά αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο εμεί ω χώρα, ω κράτο μέλο, προτείναμε χαμηλότερο αριθμό γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε βαθμιδών και αν. Ε, ε, λειτουργήσει ή δεν λειτουργήσει την πρώτη φορά, μετά θα προτείνουμε και άλλους. Ε, οι δυνατότητες μετεγκατάσταση και όλη μετεγκατάσταση σε μια εβδομάδα, ε, τι κάναμε, δεν έχουμε hot spot, απλώς μεταφέρουμε ανθρώπους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα σε αυτές τις εγκαταστάσεις υποδοχής, ε, να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής και να γίνεται σοβαρή δουλειά όχι απλώς ε, να είναι μια παράσταση και να λέμε ότι τους μεταφέραμε, τους βάλαμε σε ένα αεροπλάνο και μετά να παριστάνουμε ότι κάναμε αυτό το οποίο μας ανηλυγεί, αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Το χρονοδιάγραμμα είναι μια διαδικασία εν εξελίξη. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε την εξέλιξη και απλώς να διασφαλίζουμε ότι προσφέρουμε τη βοήθεια που απαιτείται. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Θέλετε να τελειώσετε στις 5, αλλά δεν ξέρω ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν θέλετε να τελειώσετε εσείς τι 5. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο συγκεκριμένο για ερωτήσεις οι οποίες ετέθηκαν. Ε, αν θέλετε να απαντήσετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, οι περισσότερες αφορούσαν αυτά τα θέματα. Οπότε νομίζω τα κάλυψα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ για την επιπλέον πληροφόρηση που μας προσφέρατε. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας ως Υπουργοί με τις ομάδες σας. Κύριος Γκιντεόν. Ένα ζήτημα που αφορά το καλέ και ακούστηκε και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο. Καλέ και Δουνκέρκη. Δεν δόθηκε απάντηση. Ναι, ασφαλώς θα θέλει να απαντήσει ο Υπουργός, παρακαλώ. είναι μάλλον πολυμερές ζήτημα, παρά ζήτημα που αφορά καθαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάνει επαφές, εγώ και από την Ολλανδική εμπειρία ξέρω ότι υπάρχουν επαφές με Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο για τη μεταφορά από το Βέλγιο και τις κατοχώρες προς το Ηνωμένο Βασίλειο και παρακολουθείτε στενά αυτό το ζήτημα. Σε σχέση με το Καλέ Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχει μικρές διαστάσεις εκεί και πολύ μεγαλύτερες στην, ε, δυτική, στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο σύστημα του ασύλου χωρίς να θέλουν να βρίσκονται εκεί και δεν προβλεπόταν αυτό νομίζω, στο συγκεκριμένο δηλαδή τόπο. Ε, και νομίζω ότι αυτό δεν το προέβλεπαν οι αρχικοί κανόνες. Από την άλλη αυτό αφήνει ένα κενό, γιατί όταν κάποιος προσπαθεί να φύγει από κάπου για να σωθεί, ζητάει άσυλο και το άσυλο σημαίνει ότι κάπου πρέπει να πάει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή ότι αυτοί που ζουν άσυλο, όσοι δεν θέλουν άσυλο στη Γαλλία για κάποιους λόγους, ή, ε, αλλιώς, πρέπει να, ε, ή αλλιώς ξέρουμε ότι κινδυνεύουν να ε, αντιμετωπίσουν μια απόρριψη της αιτήσεώς τους. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί πρέπει να βλύσεις ε, στο πρόβλημα, να τις υποστηρίξουμε στο βαθμό του δυνατού γιατί είναι και οικονομικό ζήτημα. αλλά δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, ξεπερνά τη συζητήσει, τη δυνατότητα για επίλυση μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ των δύο εμπλεκομένων χωρών. Ε, προχωράει καλά, υπάρχουν ε, πολλές συζητήσεις, πολλές προόδοι έχουν σημειωθεί και έτσι αν τυχόν προκύψουν ε, νέες δυσκολίες, αν αυξηθούν οι αριθμοί, θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε ίσως. Πάντως προς το παρόν εμείς ως κράτος μέλος είμαστε εμπλεκόμενη πλευρά. Αλλά δεν είναι ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει το Συμβούλιο στην πλήρη σύνθεσή του. Γι' αυτό ως Προεδρία είναι δύσκολο να σχολιάσω. Ο Πρόεδρος. Πιστεύω κύριε Υπουργέ ότι βλέπετε ποιε είναι οι προτεραιότητες μας εδώ από τι τοποθετήσει των συναδέλφων. Τα γνωρίζουν καλά τα θέματα, όλοι έχουν εμπειρία. Είναι ζητήματα σχετικά και με τη μετανάστευση που μας απασχολούν. Επιταχύνουμε και εμεί στο κοινοβούλιο τη εργασία μας. του κυρίους Δε Ιόγκ και Κάλλη νομίζω βλέπετε πώς βλέπουμε την ε, κατάσταση. Ο κύριος Κύρκος αναφέρθηκε στην Ελλάδα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται και στα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αίσθηση ότι αντιμετωπίζουμε μια πραγματική κρίση και ότι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να δοθούν λύσεις και απαντήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν μια πολύ λεπτομερή επικοινωνία μαζί σας ε, εβδομαδιαία βάση για τα θέματα αυτά. Και ασφαλώς και στα νομοθετικά ζητήματα θα υπάρξει εντατική συνεργασία όπως είχαμε και με την προηγούμενη Προεδρία. Αλλά βλέπω, νομίζω, βλέπετε νομίζω ότι έχουμε πολλά θέματα για την επανεγκατάσταση, για όλα αυτά τα ζητήματα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα στο Σέγγεν. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν που ήρθατε. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να σας ξαναδούμε. Και αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την υπομονή σας, την παρουσία σας εδώ. Η επόμενη συνεδρία στις 14 Ιανουαρίου, πέμπτη δηλαδή, αυτής της εβδομάδας. Πάντως, πάντως σημειώνω πως κοιτάμε στο δυνατόν να μην γίνεται συνεδρίαση μέσα στην ίδια εβδομάδα Δευτέρα και Πέμπτη. Ελπίζω να με ακούσατε όλοι. Είπαμε ότι δεν θα κάνουμε συνεδριάσεις μέσα στην ίδια εβδομάδα Δευτέρα και Πέμπτη, εκτός και ένα απολύτως απαραίτητο. Για δε τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο, ζητώ συγγνώμη. Και θα ε, φροντίσουμε σε επόμενη συνεδρία.